Dear colleagues, welcome to the afternoon session. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε. Έχουμε δημόσια κρόση και θα παρακολουθήσουμε πρώτα απ' όλα την παρουσίαση των συμπερασμάτων μας από την επίσκεψη που κάναμε στην Βιέννη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταρχήν, πρόκειτο σήμερα το πρωί να παρουσιαστεί αυτή η έκθεση, αλλά επειδή έγιναν κάποιες αλλαγές στην ημερήσια διάταξη, αναγκαστήκαμε να το αλλάξουμε. Ο κύριος ε, Νάγκη, λοιπόν, θα μας ε, ενημερώσει τα αποτελέσματα, για τα αποτελέσματα της επίσκεψης αυτής. Παρακαλώ κύριε Νάγκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όντω πριν από δύο εβδομάδες είχαμε μια πολύ ευχάριστη επίσκεψη στην Βιέννη. Συμμετείχαν η κυρία Τσίνικη, ο Φρανς Βέκα και προσωπικό από την Επιτροπή μας. Μας παρουσιάστηκε το έργο λοιπόν του οργανισμού αυτού, το πλαίσιο μέσα στο οποίο δουλεύει και ποια είναι τα τμήματα του οργανισμού. Μάθαμε για τους τρόπους με τους οποίους εργάζονται, για τις έρευνες που κάνουν και επίσης μας κάλεσαν και καλό και εγώ όλους τους συναδέρφους στο φόρουμ που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πήραμε και πληροφορίες για την υπηρεσία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το έργο της στην Ελλάδα, στα hot spots. Συναντηθήκαμε και με διάφορους φορείς, αξιωματούχους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ινστιτούτα και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το ΦΡΕ ετοιμάζει μια έκθεση, ο οργανισμός δηλαδή αυτός για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδική έκθεση όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση και θα συζητηθεί λεπτομερέστερα στο φόρουμ που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, όπως είπαμε. Η αντιπροσωπεία υπογράμμισε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τον ρόλο και των μη οργανώσεων αλλά και των εθνικών κοινοβουλίων προκειμένου να υπάρχει καλή συνεργασία υπογραμμίζουμε ότι υπάρχουν καλές πρακτικές σε χώρες μέλη και ότι θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή τέτοιων βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε θέματα όπως η πρόσφατη μεταναστευτική κρίση. Για να προστατεύσουμε μεταξύ άλλων τα παιδιά. Ε, χρειάζεται επίσης να έχουμε και έρευνες καλού επίπεδου και εκθέσεις καλού επίπεδου, ώστε να μπορούμε να συλλέξουμε αξιόπιστα στοιχεία για το έργο μας. Ζητήσαμε λοιπόν από το ΕΦ από τον οργανισμό να μας προσφέρει ειδικέ εκθέσεις και ειδική βοήθεια για το δικό μας το έργο. Αυτά με δύο λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, παρακαλώ, εσείς που συμμετείχατε στην αντιπροσωπεία, ο Τσίνσκι πρώτα, παρακαλώ. Η κυρία Κινίτσι, ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι όντω συμμετείχα στην αποστολή στην Βιέννη, στη συνάντηση με τον Φρά και συμφωνώ πολύ με όσα είπε ο επικεφαλή τη επισκεψή μα, ο συνάδελφος, Να υπογραμμίσω ότι στη συνάντηση που είχαμε στα γραφεία της ΦΡΑ μάθαμε τη δουλειά που κάνει ο οργανισμός αυτός στο επίπεδο της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τις έρευνες, τις ανακρίσεις, τις συνεντεύξεις μέσω των οποίων συγκεντρώνει αποτελέσματα, τα πορίσματα στα οποία καταλήγει και τη συμβολή όλης αυτής της δουλειάς για τις κυβερνήσεις σε εθνικό επίπεδο και για να μας εκπροσωπήσει βεβαίως στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θίξαμε διάφορα θέματα όπως την όπως αν και με πρόλαβε ο συνάδελφος, ένα αποτέλεσμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του φαινομένου της μετανάστευσης. Ένα φαινόμενο εξαιρετικά περίπλοκο, το οποίο νομίζω μια από τις κρίσιμες στιγμές είναι ακριβώς η προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων που είναι αναγκασμένοι να καταλέψουν τις αιστείες τους και στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Αυτό πραγματικά με έκανε να θαυμάσω το, τη δουλειά του Φρά είναι ότι πολύ γρήγορα ο Φρά έχει αποστείλει εμπειρογνώμονες και ειδικού στην ε, Ελλάδα ως αποσπασμένους υπαλλήλου. Ήταν σημαντικό αυτό και είναι πολύ σημαντικό κυρίως για την προστασία των μεταναστών και ιδίως των ανηλίκων. Αυτή η τελευταία ενέργεια του ΦΡΑ έχει διπλή αξία. Πρώτον, ότι δίνει πραγματική υλική στήριξη στα κράτη-μέλη και από την άλλη μαρτυρά την ανάγκη να ελέγχουμε και να απαλληθεύουμε το κατά πόσον τα δικαιώματα των μεταναστών προστατεύονται επαρκώς. Και βεβαίως να διεκδικούμε να γίνονται σεβαστά αυτά. θα ήταν καλό να δημιουργηθεί και ένα εγχειρίδιο από τον ΦΡΑ για του υπαλλήλου όσων ασχολούνται με τα θέματα του ασύλου και εξετάζουν τι σχετικέ αιτήσει. Υπάρχει μια σχετική προσπάθεια και μου φαίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό. Και κάτι που είχα πει ήδη από τον Γενάρη για τους αλλοδαπού ε, ασυνόδευτού ανηλίκου να γίνει μια μελέτη δείγματος και αυτό βάσει ενός χεριδίου με ε, συστάσεις για το τι πρέπει να προσέχει κανείς ε, στην προσπάθεια προστασίας των ε, μεταναστών, ιδίως των πλέον ευάλωτων, δηλαδή των ανηλίκων. Μια τέτοια προσπάθεια θα μας βοηθήσει γενικότερα να πλαισιώσουμε σωστά το φαινόμενο της μετανάστευσης και θα διευκολύνει τις δικές μας δράσεις και όσων καλούνται να αναλάβουν δράσεις στα πλαίσια της μετανάστευσης. Η επίσκεψή μας λοιπόν νομίζω επιβεβαίωσε την ανάγκη να συνεχίσει το σημαντικό, της έργο, το σημαντικό του έργο οργανισμός και υπογράμμισε την ανάγκη εμείς ως Κοινοβούλιο, όλος ιδιαίτερος αλλά και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, να αξιοποιήσουμε τη συμβολή του οργανισμού ΦΡΑ. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι οι συστάσεις σας, σε συνδυασμό με τις συστάσεις του κυρίου Νάγκη, θα είναι πολύ χρήσιμες για την μελλοντική συζήτηση. Τώρα Κυρίες και κύριοι ομιλητές, αγαπητοί ευρωβουλευτές, είναι χαρά μου που σας καλωσορίζω σε αυτήν εδώ την ακρόαση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 εκ μέρους του κυρίου Κλοντ Μωράης, ο οποίος μου ζήτησε ως, ε, αντιπροέ... ως αντιπρόεδρο της Επιτροπής Λίμπε να τον εκπροσωπήσω σήμερα το απόγευμα. Έχει πλέον γίνει παράδοση για τη Λίμπε να οργανώνει αυτή την ακρόαση που ε, πλαισιώνει τις εργασίες μας ε, για την ετήσια έκθεση όσον αφορά την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με μεγάλη μας χαρά καλωσορίζουμε τους εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων για να παρουσιάσουν στους Ευρωβουλευτές την εργασία που έχει γίνει σε αυτό το τομέα. Στο ψήφισμα της 8 η Σεπτεμβρίου 2015 για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε ότι είναι απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά της όργανα και τα κράτη-μέλη να εγγυηθούν τον σεβασμό και την πρόθεση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών που εγγράφονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό θα πρέπει να γίνει ε, στην ευρωπαϊκή και στην ε, εθνική νομοθεσία, στις δημόσιες πολιτικές και κατά την εφαρμογή τους και θα πρέπει πάντοτε να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας. Με χαρά μου δίνω το λόγο στον κύριο Νάγκη και πάλι για να κάνει κάποια εισαγωγικά σχόλια. Κύριε Νάγκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ως ε, εισηγητής της έκθεσης για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος, ε, με χαρά μου βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτήν εδώ την ακρόαση έτσι ώστε να συμμετάσχω σε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά στην καθημερινή μας ζωή και μας προστατεύουν ως άτομα αλλά και ως μέλη ομάδων. Κανείς εξ η οποία ενδεχομένως να χρειαστεί μια τέτοια μορφής προστασία. Ε, μπορεί να ανήκει σε κάποια μειονότητα που να χρειάζεται την προστασία του νόμου. Τα δικαιώματα αυτά λοιπόν είναι εγγυημένα από τον νόμο, όμως πολλές φορές δεν εφαρμόζονται. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατή ευκαιρία για να τονίσουμε τη σημασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να θεωρεί τον εαυτό της ηγέτη στον κόσμο όσον αφορά στα δεμελιώδη δικαιώματα, θα πρέπει να γνωρίζουμε καταρχάς πώς είναι η κατάσταση εντός της Ευρώπης. Και ε, οι χώρες ε, που ε, θέλουν να μπουν στην Ένωση, και αυτές είναι ε, κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε, γιατί και η κατάσταση εκεί πολλές φορές είναι προβληματική. Πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, ε, καθώς οι απαιτήσει εκεί ε, μπορεί να είναι μεγαλύτερες από ό,τι στις δικές μας χώρες. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε σήμερα να μιλήσουμε για διάφορα ζητήματα, για τους Ρωμά, για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ, για τους ανθρώπους με αναπηρία. Εγώ επίσης ανήκω σε μια εθνική μειονότητα. 40 ε, εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ανήκουν στις εθνικές μειονότητες. Μάλιστα έχουμε εδώ ε, ομιλητή, ο οποίος θα μιλήσει για την κατάσταση μιας εθνικής μειονότητας. Τα τελευταία χρόνια αυτό το θέμα έχει κερδίσει το ενδιαφέρον και αποκτά και μεγαλύτερη σημασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς ε, ε, όλο και περισσότερο μιλούμε επικοδομητικά για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Νομίζω ότι και εδώ και στην έκθεση μπορούμε να ε, στηρίξουμε τέτοια ζητήματα. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ για να ακούσω τις παρουσιάσεις σας. Ευχαριστούμε για τη σύντομη παρουσίασή σας. Τώρα θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας ε, και στο τέλος κάθε μίας εκ των δύο συνεδριών θα υπάρξουν ερωταπαντήσεις. Παρακαλώ να ξέρετε ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο αυτή η συνεδρίαση και θα καταγραφούν και οι παρεμβάσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη συνεδρία, τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015, αξιολόγηση των επιτευγμάτων και των προκλήσεων. Θα ξεκινήσουμε τώρα με το πρώτο πάνελ. Έχω τη χαρά να καλωσορίσω τον κύριο Φραντσέσκο Φωνσέκα Μορίλο, ε, υποδιευθυντή, ε, γενικό υποδιευθυντή για την ε, δικαιοσύνη και τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα εκπροσωπήσει τον κύριο Τίμερμανς που είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας. Ε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντα τη συγνώμη του πρώτου αντιπροέδρου, ο οποίο τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να συνδυάσει τι ηλυμένε του υποχρεώσει με την παρουσία του εδώ. Είναι οι Ευρωπαϊκέ Μέρε Ανάπτυξη έτσι κι αλλιώ και άλλαξαν ε, οι ώρες του ραντεβού, το ραντεβού με τους Αφρικανούς Υπουργούς. Ε, γι' αυτό ε, μου είπε να έρθω στη θέση του να τον εκπροσωπήσω και σας ζητά συγγνώμη πάνω από όλα βεβαίω την αντικατάσταση αυτή μου ζήτησε να σα μεταφέρω το μήνυμα, το μήνυμα που ο πρώτο αντιπρόεδρο θα ήθελε να σας ε, μεταφέρει ο ίδιος με την αφορμή αυτή τη ακρόαση. Κυρίε και κύριοι, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Έχει δημιουργηθεί οργή λόγω της χρηματοπιστωτική κρίσης ε, και οι εργαζόμενοι πολίτες έχουν ήδη πολλά προβλήματα. Η μετανάστες έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των μεταναστών. Οι πρόσφατες επιθέσεις στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες είναι μία πραγματική απειλή ε, των φόντα μεταλλιστών κατά των βασικών αξιών του τρόπου ζωής μας. Οι φόβοι των απλών πολιτών είναι ότι θα τους κατακλείσουν πρόσφυγες, ότι θα ισλαμοποιηθεί η Ευρώπη, θα εξισλαμιστεί δηλαδή. Φόβος για την χρηματοπιστωτική κρίση, ότι θα γλιστρήσουν στη φτώχεια της οικονομικής κρίσης, ότι θα τους επιτεθούν τρομοκράτες. Φόβος με τον ένα τον άλλο τρόπο. Όταν ο φόβος κυριαρχεί, βλέπουμε μόνο τις απειλές και όχι τις ευκαιρίες. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτού του φόβου και να αναζητήσουμε συνομιλητή στο πρόσωπο του άλλου. Και εκείνο έχει μια ιστορία να αφηγηθεί και ίσως και το συμφέρον ε, ε, προσφέρει σε μια κοινωνία που βασίζεται σε κοινέ αξίε όπω η ανεκτικότητα, η δημοκρατία, η αλληλεπίδραση και ο αμοιβαίο σεβασμό. Στην έκθεσή μα για την υλοποίηση τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχουμε προβλέψει ιδιαίτερο κεφάλαιο που σκοπό έχει μαζί με την ετήσια ημερίδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα να οργανώσει συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα εναλλακτική προς όσα επικρατούν και λέγονται με πηγή το φόβο. Η έκθεσή μας για την ετήσια χάρτα περιλαμβάνει ακριβώς αυτή την ειδική σύνοδο που οργανώθηκε στην πρώτη ημερίδα τον περασμένο Οκτώβριο με θέμα την ανοχή και το σεβασμό προλαμβάνοντας και ε, διαλύοντας τις αντισημιτικές και αντιισλαμικές τάσεις στην Ευρώπη. Εθνικοί και Ευρωπαίοι πολιτικοί ηθήνοντες, πρόσωποι της διεθνούς και ε, τοπικής ε, κοινωνίας των πολιτών, συζήτησαν σε αυτή τη σύνοδο για τους λόγους τα γενεσιουργά αίτια του κλίματος κατά των ε, Εβραίων και Ισλαμιστών στην Ευρώπη. Ε, αναλύσαμε τις σημερινές τάσεις και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να αναχαιτήσουμε το μίσος και να ε, καλλιεργήσουμε ένα πολιτισμό ανοπτικότητας. Η ημερίδα μας αυτή κατέληξε σε μια συγκεκριμένη σειρά από πράξεις οι οποίες ε, ήταν, ε, ένα, ε, ήταν το αντικείμενο του ειδικού κεφαλαίου της έκθεσής μας, μια από τις βασικές δράσεις που αναλύθηκε που αναγράφεται στο κεφάλαιο αυτό της έκθεσης είναι η αιτήσια συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εταιρείες πληροφορικής, εκπροσώπους των κρατών μελών και της κοινωνίας των πολιτών για να αντιμετωπίσουν αυτήν την λογική μίσους που έχει επικρατήσει. Η τελευταία ε, σύνοδος ήταν στι 31 Μαΐου με τη δημοσίευση ενός κώδικα διοντολογία. Οι εταιρείες πληροφορικής όπως ε, το Google, το Twitter, το Facebook, η Microsoft συμφώνησαν να αποτιμήσουν το περιεχόμενο που έχει εκφράσει μίσου. Ε, αντίθετα με το εθνικό μας δίκαιο και ε, εφαρμόζοντα την Ευρωπαϊκή Απόφαση για τον Ρατσισμό και την Ξενοφόβια. και βάσει των διεθνών προποθέσεων. Εάν προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία, το επιγραμμικό περιεχόμενο με εκφράσει μίσου θα ε, καταργείται από το διαδίκτυο εντό 24, 24 ώρων. Πρέπει να προσπαθήσουμε όμω ε, και εκτό διαδικτύου προ την ίδια κατεύθυνση. Πρέπει να μην επιτρέψουμε να δημιουργούνται αιστείε αντισημιτισμού και αντιισλαμισμού που να παροτρύνουν στην βία. Πρέπει η αστυνομική και η εισαγγελική αρχή κάθε χώρας να μπορεί να στηρίζει και να δίνει ε, τις δυνατότητες στην κοινωνία των πολιτών να αναπτύξουν και τις αντίθετες ε, λογικές και εκφράσεις. Οι, εταιρείε πληροφορικής πρέπει να καλλιεργήσουν την ελευθερία έκφρασης αλλά δεν είναι μέρος αυτής η έκφραση μίσους. Οι διάφορες πρωτοβουλίες για την καλλιέργεια διαλόγου και ανταλλαγών καθώς και πιστές τις μέτρων για να καταπολεμήσουμε τον ρατσισμό και την ξενοφοβία στην ε, κοινωνία υποδοχής είναι ε, τα μέσα για να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο κλίμα ώστε να αντιμετωπίσουμε το τοξικό κλίμα γύρω από τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που καλλιεργούν απλώς προκαταλήψεις και φόβους στον πληθυσμό αλλά και πραγματικό μίσος οι σωματικές και λεκτικές επιθέσεις κατά των προσφύγων και μεταναστών ή κατά των όσων γίνονται αντιληπτοί ως ξένοι έχουν ενταθεί σε πολλά κρατημέλη. Είναι μια ανησυχητική τάση που χαρακτηρίζεται από τι αντιμουσουλμανικές κυρίως τάσεις. Οι εκφράσει ρατσισμού και ξενοφοβία πρέπει να γίνουν προτεραιότητα για μα ω προ την καταπολέμησή του. Απαιτούν κοινέ προσπάθειε. Ξέρουμε ότι οι νόμοι είναι καλοί μόνο αν εφαρμόζονται πραγματικά. Εργάζομαι εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να στηρίξω την ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου, την διακομματική ομάδα κατά της, ε, ε, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα μια νέα πλατφόρμα για ανταλλαγές με όσους ασχολούνται με την χάραξη πολιτικών κατά του ρατσισμού και της ε, ξενοφοβίας, ώστε να συνδυαστούν οι προσπάθειες κατών μελών, κοινωνίας των πολιτών και άλλων διεθνών οργανισμών. Ήθελα να τονίσω τον πολύ θετικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΦΡΑ ο Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στη Βιέννη. Να πω ότι πρέπει να υπάρξουν στοχευμένες δράσεις ε, και ε, με στοχευμένη χρηματοδότηση για να πετύχουμε τους σκοπούς μας. Ε, μια άλλη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα άλλο κεφάλαιο τη ετήσια έκθεσης. Το 2015 με το πακέτο για την καλύτερη νομοθεσία, το καλύτερο νομοθετήν, επιβεβαιώσαμε την αρχή ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν ένα απόσπαστο μέρο τη διαδικασία μελετών αντικτύπου. Η συμφωνία για, την, για το καλύτερο νομοθετή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την ενίσχυση τη συμμόρφωση με τι υποχρεώσει για τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσω αυτή τη διαδικασία. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα υποχρεώνται να λάβουν υπόψη την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλε του τι δράσει, όχι μόνο στα νομοθετικά του μέτρα. Αυτό συμπεριλαμβάνει την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και τη σύναψη διεθνών συμφωνιών το 2015 λόγω χάρη με εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές ε, ε, απαιτήσαμε να λαμβάνονται υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και στη σύναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Η απόκριση που είχαμε δείχνει ότι δεν μπορούμε να ε, συμβιβαστούμε με μερικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν προτείνουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και για να πετύχουμε ένα χώρο ελευθερία, δικαιοσύνη και ασφάλεια κοινό, πρέπει να αναλάβουμε και κοινή δράση για να προωθήσουμε και να αυξήσουμε τον πύχη ω προ το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Σε αυτό το πλαίσιο, το πακέτο για τη μεταρρύθμιση ε, των ε, νομικών μέτρων, όπω το τεκμήριο αθωότητα ή τη παρουσία σε μια δίκη ή των ε, ειδικών μέτρων για την παρουσία παιδιών ανηλίκων σε ποινικέ διαδικασίε, θα εκπροσωπήσει το πρώτο σκέλο τη αλλαγή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά ολοκληρώθηκαν πρόσφατο χρονικό διάστημα. Τώρα πρέπει να παρακολουθήσουμε την υλοποίηση των μέτρων αυτών. Η έκθεση επίσης δείχνει πώς εφαρμόστηκε η χάρτα και στα κράτη-μέλη και από τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι αυξάνεται η σημασία της διαδικασίας που παραβάσει και το πώς, ε, πώς ανατρέχουμε σε αυτές. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα κράτη-μέλη ανατρέ... Ε, σέβονται την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων όταν εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου 2015 ξεκινήσαμε 49 διαδικασίες επί παραβάση κατά κρατών μελών για την ε, πλημελή υλοποίηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Η εικόνα και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο δεν είναι πάντοτε φωτεινή και ευχάριστη. Ε, το 2015 ήταν δύσκολη χρονιά για τα θεμελιώδη δικαιώματα, κυρίως λόγω των διαφόρων μορφών κρίσης που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Ε, πιο σημαντικό από ποτέ είναι να βεβαιωθούμε ότι οι νόμοι δράσεις μας και ε, πολιτικές μας ε, διέπονται από τις κοινέ μας αξίες και πρέπει να αναζητήσουμε την, τον πλήρη σεβασμό της Χάρτας των Θεμελιδών Δικαιωμάτων. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ πολύ σύντομα στο μέλλον. Ε, 17 και 18 Νοεμβρίου του 2016 θα έχουμε την επόμενη ημερίδα για το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Κατά αυτόν. Στο άρθρο 11 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναφέρονται η ελευθεροτυπία και η ελεύθερη έκφραση, βασικές θεμελιώδεις αξίες από τον οποίο βασίζεται η Ένωση. Η ημερίδα θα διερευνήσει τις διασυνδέσεις μεταξύ ελεύθερων και πολυφων, πολυφωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τη μια και τη σχέση τους με τη δημοκρατία την άλλη. Δημόσιες διαβουλεύσεις ε, γύρω από την ημερίδα ήδη ξεκίνησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την 1η ως την 14η Ιουλίου ε, θα γίνουν οι ε, καθεαυτές συζητήσεις. Καλό όλους να συμμετάσχουν για να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο πλαίσιο ώστε να έχουμε μια πρόσφορη συζήτηση. Παρακαλώ να συμμετάσχετε ε, στο βαθμό που είναι δυνατό στην ερχόμενη ημερίδα. Και επίση να σας πω ότι τα συμπεράσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Παρακαλώ να συνεχίσετε κι εσείς να τα προωθείτε και να τονίζετε την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου ανά την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very Ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Πολ Φανσάσε Φανάισελτ και τον κύριο Μαρτέιν Ντεγράδα που εκπροσωπούν την Ολλανδική Προεδρία συμπροεδρεύουν τη ομάδα εργασία για τα θεμελιώδη δικαιώματα, δικαιώματα των πολιτών και ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, των ΦΡΕΜ. Ε, κύριε Πολ ε, Φανσάς Φανέισελτ και κύριε Μαρτέιν Τιγράβε έχετε το λόγο για ένα τέταρτο περίπου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Εξότιμοι ευρωβουλευτές και άλλοι προσκεκλημένοι εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν πολύ που μας καλέσατε ως πρόεδροι της ΦΡΕΜΠ, της ομάδας εργασίας δηλαδή του Συμβουλίου που ασχολείται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτη και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Με μεγάλη χαρά λοιπόν και είναι και τιμή μας εξάλλου να σας παρουσιάσουμε τις δραστηριότητές μας κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας. Θα αρχίσουμε το δεύτερο ετήσιο διάλογο για το κράτος δικαίου στο Συμβούλιο. Με την τελική Προεδρία το Συμβούλιο κατέληξε συμπεράσματα τα οποία ζητούσαν από το Συμβούλιο να βρει ένα πλαίσιο για να συζητήσει τα θέματα κράτου δικαίου. Και το Συμβούλιο είχε τον πρώτο ετήσιο τέτοιο διάλογο τον Νοέμβριο που μα πέρασε υπό την Προεδρία του Λουξεμβούργου. Η Προεδρία των Κατόχωρων λοιπόν οργάνωσε μια δεύτερη συζήτηση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων το μήνα που μας πέρασε. Το θέμα ήταν η πρόκληση να διατηρήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες μεταξύ άλλων και το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα όταν ε, εντάσσουμε στις κοινωνίες μας πρόσφυγες και μετανάστες. Ακολούθησε και ένα σεμινάριο με το ίδιο θέμα στο Στρασβούργο που οργάνωσε η Προεδρία σε συνεργασία με το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Ε, στο διάλογο είχαμε εισαγωγή από τον Διευθυντή της ε, Υπηρεσία Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τον κύριο Μάικλ Φλάχερτη. Ο διάλογος ήταν ανοιχτός, η συζήτηση ήταν, έγινε με ειλικρίνεια και με συμμετοχή πολλών χωρών μελών. Η συζήτηση έδειξε ότι πολλές χώρες μέλη αντιμετωπίζουν αντίστοιχες προκλήσεις. Η ένταξη είναι βέβαια εθνική αρμοδιότητα, αλλά από την άλλη μεριά Ό,τι συμβαίνει σε μια χώρα έχει επιπτώσει σε μια άλλη χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, όλε οι χώρε μέλη είναι υποχρεωμένε να σέβονται τα ίδια διεθνή στάνταρτ. Συγχρόνω δεν μπορούμε να πούμε ότι μία λύση ταιριάζει σε όλου όταν πρόκειται για ένταξη. Οι χώρε μέλη λοιπόν ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικέ και προτάσει. Και Τέτοια συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου και στο πρόγραμμα δράση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έλαβε υπόψη τη. Επιτρέψτε μου εδώ να σα πω ότι και κατά την προετοιμασία του διαλόγου αυτού ε, υποφελθήκαμε πάρα πολύ από τι συνομιλίε που είχαμε με πολλές ε, οργανώσεις τη κοινωνία των πολιτών. Ο διάλογο για το Κράτο δικαίου λοιπόν θα αξιολογηθεί στο Συμβούλιο πριν από τα τέλη τη χρονιά αυτή. Και ελπίζουμε ότι δύο διάλογοι που έλαβαν χώρα μέχρι τώρα έδειξαν την πρόσθετη αξία τέτοιων συζητήσεων για το κράτος δικαίου και ότι καλό θα ήταν να γίνονται τακτικά στο Συμβούλιο. Επιτρέψτε να αναφέρω εδώ και την, το έργο μας όσον αφορά την ε, ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπως ε, είπα, εκ μέρους του Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της ακρόασης για το θέμα αυτό, στις 14 Απριλίου, το Συμβούλιο τόνισε ότι θέλει να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας επίσης κάναμε και περισσότερα πράγματα σε θέματα τεχνικού χαρακτήρα ή διαδικαστικού που έχει θέσει μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Συμβούλιο λοιπόν περιμένει τώρα την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις επιλογές τις οποίες θα καταλήξει για να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η συνεργασία μας στον τομέα της ΚΕΠΑ. Δύο θέματα δηλαδή που έχουν καθοριστεί σαν πολύ ευαίσθητα. Ε, το Συμβούλιο θα εξετάσει την ανάλυση αυτή και θα προχωρήσει επί Σλοβακικής Προεδρίας. Από την πλευρά μου θα ήθελα επίσης να αναφέρω την πρόταση της Επιτροπής για την πρόσβαση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Σύμβαση για την ε, πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την ενδοικογενειακή βία που ονομάζεται Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε αφιερώσει πάρα πολλές συναντήσεις και πολλή δουλειά και ελπίζουμε θα συνεχιστεί με την επόμενη Προεδρία. Και τώρα επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να δώσω το λόγο στον Συνπρόεδρο, τον Πολ Σάσεφανέισελτ. Ευχαριστώ πολύ, Μαρτέν, και ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και για μένα είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ για να σα ενημερώσω για τι δραστηριότητέ μα όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά τη διάρκεια τη Ολλανδική Προεδρία. Κυρίω θέλω να επιστήσω την προσοχή σα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατά το έτος 2015, συμπεράσματα τα οποία έκρινε το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων την Πέμπτη μας πέρασε στις 9 Ιουνίου και θέλω να σας ενημερώσω και τις σχετικές δραστηριότητε μας για να καταλήξουμε εκεί. Πρώτον, θέλω να αναφερθώ σε αυτό εδώ το βιβλιαράκι που μιλάει για στιγμές μιζέριας και καταστροφών. Και θα ήταν ίσως καλό να το έχουμε όλοι υπόψη μας αυτή την εποχή και γράφτηκε το 1584 από τον Γιούστιους Λίψιους. Το όνομα αυτό το γνωρίζετε βέβαια όλοι πολύ καλά γιατί είναι το όνομα του κτηρίου που συνεδριάζει το Συμβούλιο. Το κεντρικό μήνυμα λοιπόν στο βιβλίο αυτό είναι ότι πρέπει να έχουμε μια στοική στάση. Και είναι πολύ χρήσιμο για μας που είμαστε συμπρόεδροι της ΦΡΕΜΠ, αλλά και όχι μόνο, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη και τα θεσμικά της όργανα της ημερών ημέρα. Αν μη τι άλλο, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο 1584 και τώρα. Και αυτή είναι ότι η κοινωνία μας, στην κοινωνία μας επικρατεί το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και γι' αυτό και έχουμε εγκρίνει διάφορα σημαντικά έγγραφα όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και έρχομαι τώρα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και το περιεχόμενό του. Θα αναφερθώ στα τρία του στοιχεία. Πρώτον, η χάρτα αυτή καθ' αυτή. Στις 19 Φεβρουαρίου η Προεδρία των Κάτω Χωρών οργάνωσε ένα σεμινάριο εμπειρογνωμόνων όσον αφορά το πώς εφαρμόζεται στο, στο εσωτερικό η χάρτα θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων. Το σεμινάριο αυτό έγινε στο Άμστερνταμ. Να δούμε δηλαδή πώς χρησιμοποιείται τη χάρτα αυτή κάθε φορά που εκπονείται πολιτική ή παίρνονται πολιτικές αποφάσεις συμμετείχαν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες μέλη και άλλοι φορείς οι οποίοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο ασχολούνται με τη χάρτα. Και κατάληξε το σεμινάριο σε διάφορα συμπεράσματα που συμπεριλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Πρώτον, δεν θα πρέπει να βλέπουμε τη χάρτα αυτή μεμονωμένα. Πρέπει να την βλέπουμε και να την εφαρμόζουμε παράλληλα με άλλε πηγέ θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεύτερον, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην διατύπωση του άρθρου 51 τη χάρτα. Και να προσέξουμε και τις διατάξεις της ε, χάρτας ε, που η ερμηνεία τους ε, δεν ευθυγραμμίζεται πάντα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τρίτον, να δώσουμε σημασία σε κατάρτιση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη χάρτα αυτή και τέλος να ζητήσουμε από τον οργανισμό να χαρτογραφήσει μελέτες και πρακτικές όσον αφορά την εφαρμογή της χάρτας στην πράξη. Δεύτερον, Πρόκειται για την συνοχή ανάμεσα στην πολιτική που ακολουθούμε στο εξωτερικό και στο εξωτερικό όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και ο κύριος Νάγκη αναφέρθηκε σε αυτό. Εδώ πέρα δεν πρόκειται μόνο να κάνουμε τα λόγια πράξη, πρόκειται επίσης και για το να μιλάμε για αυτά τα οποία κάνουμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τρόπους συνεργασίας. Το Μάρτιο το ΦΡΕΜΠ είχε κοινή συνάντηση με το COHOM, την ομάδα εργασίας δηλαδή που ασχολείται με τα θεμελιώδη δικαιώματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερευνητές λοιπόν από την ΦΡΕΜΠ και από τον οργανισμό αυτό συνεργάστηκαν και καταλήξαμε σε ένα έγγραφο με ερωτήσεις προς συζήτηση που οδήγησε σε μια πολύ καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων. Μεταξύ άλλων το Συμβούλιο κατέληξε να κοιτάξει καλύτερα αυτό που ονομάζουμε lines to take, το τι δηλαδή γραμμή πρέπει να ακολουθήσουμε και στα πλαίσια του COHOM και στα πλαίσια της FREMP και να είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε και σε τρίτες χώρες τι συμβαίνει εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, έχουμε ανταλλαγή απόψεων και να είμαστε συνεπείς όσον αφορά τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Και το τρίτο συμπέρασμα ήταν ότι θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία που έχει η καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Ο κ. Φονσέκα αναφέρθηκε στη σημασία του θέματος αυτού ακριβώς πριν από μένα. Στις 28 και 29 Απριλίου η Προεδρία των Κάτω Χωρών μαζί με το ΦΡΑ υποδέχτηκαν την τέταρτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την βελτίωση της αναφοράς και της καταγραφής εγκλημάτων μίσους. Εκεί ο ΦΡΑ παρουσίασε ε, τα δικά του συμπεράσματα και τις δικές του πρακτικές για την καταπολέμηση του εγκλήματος αυτού. Τα κύρια συμπεράσματα του Συμβουλίου ήταν πλήρη υποστήριξη τη νέα ομάδα υψηλού επίπεδου τη Κομισιόν για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβία και άλλων ε, φορμό, ε, μορφών αδιαλαξία. Δεύτερον, συμμετοχή τη ΦΡΑ στη νέα αυτή ομάδα για να αναπτύξουν κοινή μεθοδολογία και να μπορέσουν έτσι καλύτερα να συλλέξουν και να καταγράψουν τα εγκλήματα μίσου. Και το τρίτο στοιχείο ήταν η στήριξη στο διάλογο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εταιρείε πληροφορική για να αντιμετωπιστεί και το θέμα τη ρητορική μίσου στο διαδίκτυο. Το είπα αυτά πριν και ο κύριο Φωτσέκα Μωρίγιο. Συνοψίζω. ω Προεδρία λοιπόν θεωρούμε ότι συνεισφέραμε προκειμένου να αναλυθούν συγκεκριμένα βήματα σε τομεί που θεωρεί πολύ σημαντικού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι θέλουμε να αναγνωρίσουμε την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το προσωπικό του και του συναδέλφου από το ΦΡΑ, όπω επίση και τι πολύ ενδιαφέρουσε ανταλλαγές που είχαμε με το Δίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στου εταίρου μα το τρίο αυτό, τη Σλοβακία και τη Μάλτα δηλαδή, για τι επερχόμενε προεδρίες του. Ευχαριστώ Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Ματίας Κρούντεν, που είναι Διευθυντής Σχεδιασμού Πολιτικής στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα, η κατάσταση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Ευρώπη. Κύριε Κρούντεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να έρθω εδώ για να μιλήσω για την τρίτη ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την κατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Να επαναλάβω κάποια πράγματα που ακούσαμε ήδη προηγουμένως. Υπάρχουν κάποια λόγια που ακούστηκαν σχετικά με την πρόοδο και τη δέσμευση για πρόοδο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ε, ε, ε, ε σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, πράγματα που κάνουν πιο ισχυρή την Ευρώπη και είχαμε και ένα επιπλέον πρωτόκολλο στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της τρομοκρατίας και της μάχης κατά των ξένων μαχητών, ε, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων περιλαμβάνει και ε, την αποτελεσματική δράση εναντί αυτών που θέλουν να τα καταστρέψουν. Το Συμβούλιο της Ευρώπης. Γιατί ετοιμάζει αυτή την ετήσια έκθεση. Νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι μεταξύ άλλων που κάνει το ε, Συμβούλιο της Ευρώπης είναι και ένας διακυβερνητικός ε, οργανισμός σε 47 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και ε, στα 28 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν κοινά στάνταρ και κανόνες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Είναι δεσμευτικά τα περισσότερα προβλήματα όταν προκύπτουν σχετικά με την παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων και προκύπτουν συχνά, ε, αντιμετωπίζονται όχι ως θέμα πολιτικής διαπραγμάτευσης αλλά ως ε, αντικείμενο αξιολόγησης από μηχανισμούς ειδικού ή από ένα ε, ειδικό ε, δικαστήριο, ας πούμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από ανεξάρτητες ε, αρχές και πυρογνώμονες. Ε, είναι όλα αυτά σαν ένα ελβετικό σουγιάς. Είναι μια μεθοδολογία για να αξιολογήσουμε τα ισχυρά και αδύναμα σημεία που έχουν τα κράτη-μέλη ω προ τη δυνατότητά τους ε, να παρέχουν τη δημοκρατική ασφάλεια και να την εγγυηθούν. Είναι ένα σύστημα ε, που έχει κάθε χώρα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί σωστά. Χρησιμοποιούμε λοιπόν όλα τα πρότυπα και τους κανόνες που υπάρχουν, τα αποτελέσματα των εκθέσεων και τα ευρήματα από την ε, παρακολούθηση για να κάνουμε ακριβώς αυτό. Στην έκθεση λέγεται λεπτομερώς ακριβώς τι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη αλλά και τι δεν πρέπει να κάνουν για να μπορέσουν να εγγυηθούν ένα αποτελεσματικό, αδέκαστο ε, δικαστικό σώμα, ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μία ε, σφίζουσα κοινωνία των πολιτών και δημοκρατικά πολιτικά συστήματα, αλλά και μία κοινωνία η οποία θα τους αγκαλιάζει όλους και θα αντιστέκεται στις εξωτερικές πιέσεις. Αυτή η μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα και από άλλους. Μπορείτε να τη δανειστείτε, μπορεί κανείς να τη χρησιμοποιήσει για να αξιολογήσει την κατάσταση σε μια χώρα ή σε μια σειρά χωρών σε οποιαδήποτε από τις περιοχές που μόλις ανέφερα, σε οποιοδήποτε από τους τομείς που μόλις ανέφερα είναι ένας καλός και ανεξάρτητος αποδικημενικός τρόπος αξιολόγησης και ταυτοποίησης των προβλημάτων και των αδυναμιών. Ο δεύτερος στόχος της έκθεσης είναι φυσικά να ταυτοποιήσει τα προβλήματα αλλά και να αξιολογήσει το μέγεθός τους για να μπορέσει να κάνει μια λίστα προτεραιοτήτων. Έχουμε πέντε επιλώνες, 23 ε, ε, παραμέτρους ε, και κάποιες εκατοντάδες κριτήρια μέτρησης που μας βοηθούν να ποσοτικοποιήσουμε τα φαινόμενα που παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή. Η ποσοτικοποιημένη αξιολόγηση είναι πολύ καλή για να κάνουμε αυτήν την λίστα προτεραιοτήτων και να ετοιμάσουμε και τις δράσεις που θα μας φέρουν τις λύσεις. Όταν μιλάμε τώρα για ευρήματα, ε, δεν θα σας ε, πω ακριβώς τι λέει κάθε σημείο της έκθεσης, την έχετε στη διάθεσή σας. Υπάρχουν όμως τρία γενικά συμπεράσματα που μπορεί κανείς να αντλήσει. Καταρχάς, η κατάσταση είναι και στους πέντε πυλώνες, ε, το δικαστικό, ε, το μέσα μαζικής ενημέρωσης και ούτε καθεξής. Αυτό είναι κάτι πολύ ανησυχητικό δεν ε, ε, διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους. Ε, δεύτερον, τα προβλήματα είναι γεωγραφικά πιο διασπαρμένα από ό,τι περιμέναμε. Δεν είναι μόνο οι συνήθεις οι υποπτοί. Βέβαια, έχουμε το ίδιο μέγεθος, την ίδια βαρύτητα στα προβλήματα, αλλά υπάρχει μια τάση προς τα κάτω, δηλαδή αδυναμία των μηχανισμών μας να και όλο μεγαλύτερη αδυναμία να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τρίτο γενικό συμπέρασμα είναι ότι πολλές από τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αναφέρονται δεν μπορούν πλέον να εξηγηθούν λόγω κάποιων μεταβατικών δυσκολιών και έλλειψης εμπειρίας σε κάποιες περιπτώσεις. Φαίνεται ότι είναι οι θελημένες πολιτικές ε, που ε, ε, επί τούτο προσπαθούν να παραβιάσουν τα στάνταρ του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είπα ότι δεν θα αναλύσω όλη την έκθεση και δεν θα το κάνω, αλλά ήθελα να σας δώσω μια γεύση αυτό που είπα μόλις τώρα, όταν μιλάμε για την ελευθερία της έκθεσης, σύμφωνα με την έκθεση σχεδόν από ε, τα μισά ε, οι μισοί οργανισμοί από τα κράτη-μέλη λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένα από την προστασία έναντι των απειλών και της βίας. Επίσης, ε, δεν είναι προστατευμένοι οι δημοσιογράφοι έναντι της αυθαίρετης χρήσης της νομοθεσίας, ειδικότερα ε, κατάχρηση των νόμων για την εξύβριση και την τρομοκρατία. Σε άλλα 33 κάτι μέλη είδαμε προβλήματα με την ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την πολυφωνία και την ε, ποικιλομορφία. Δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση στα 26 από τα 35 κράτη για τα οποία έχουμε δεδομένα. Λίγο πολύ βλέπετε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση που ε, μας ε, παρουσιάζει αυτή η έκθεση. Να πω επίσης ότι η έκθεση προτείνει άμεσες λύσεις για τις καταστάσεις που διαπιστώνονται. Οι περισσότερες πρέπει να γίνουν σε επίπεδο κρατών μελών. Οι συστάσεις απευθύνονται στα κράτη-μέλη και θα περιληφθούν στα προγράμματα συνεργασίας που συχνά υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια σειρά συγκεκριμένων προτάσεων για τη δημιουργία ενός νέου Μηχανισμού για την προστασία των ανθρώπων που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα υπερασπίζονται ε, γιατί το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, θέλει να έχει συγκεκριμένα κωδικοποιημένα στάνταρ για τη μαζική παρακολούθηση την ανεξαρτησία ε, του νομικού, του δικαστικού συστήματος, ένα πρόβλημα που υπάρχει στα περισσότερα κράτη-μέλη. το τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω έχει να κάνει με το βασικό πολιτικό μήνυμα που θέλει να περάσει ο Γενικό Γραμματέα από την έκθεση και αντικατοπτρίζεται στον πλήρη τίτλο. Η κατάσταση τη δημοκρατία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη κράτου δικαίου. Είναι ένα ζήτημα ασφάλεια. Αυτή η ασφάλεια. Ε, ε, δεν ήταν, ήταν κάποτε δημοκρατική, τώρα είναι απλώς ασφαλεία γιατί θέλουμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία της σωστής λειτουργίας των οργάνων που διασφαλίζουν τη δημοκρατική ασφάλεια ε, και προσπαθούν να εγγυηθούν την ε, συνεχή και βιώσιμη ασφάλεια στις χώρες μας. Ειδικότερα ε, υπό το φως της κατάστασης που και πάλι δεν θα περιγράψω γιατί την έκανε πολύ καλά ο προλαλής σας. Στην κατάσταση λοιπόν που βρισκόμαστε σήμερα έχει αλλάξει η ταχύτητα. Βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς ανασφάλειας, το οποίο εκμεταλλεύονται όσοι θέλουν να έχουν από αυτό πολιτικά ωφέλη. Και πολύ συχνά ε, λέμε ότι το να αγγιηθεί την ασφάλεια των πολιτών ε, σημαίνει ότι τηρείς τα δημοκρατικά δικαιώματα και το κράτος δικαίου ε, εξορισμού ο Γενικός Γραμματέας ε, θέλει να στείλει το εξής μήνυμα. Με την ε, τήρηση των κοινά συμφωνημένων προτύπων και προσπαθώντας να βρούμε αποτελεσματικές και λογικές λύσεις, ε, θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε τις απειλές και να αντιμετωπίσουμε τις ανασφάλειες που προκύπτουν από το στο σύγχρονο κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Η τελευταία παρουσίαση σε αυτό το πάνελ είναι από τον καθηγητή Ολιβιέντε Σιούτερ. Κύριε είναι καθηγητής του Καθολικού Πανεπιστημίου στην Λουβέν, στο Βέλγιο και ήταν πριν συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου ανεξάρτητων ε, ειδικών όσον αφορά τα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα συζητήσει μαζί μας το θέμα της συνέχειας που δίνεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8 Σεπτεμβρίου του 2015 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μελέτη που ζητήθηκε από την ε, υπηρεσία Πολιτική όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών και στεγματικά δικαιώματα. Κάτι που ζήτησε η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ο κύριος Σιούτερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως καλύτερα να πω Αντιπρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Και είναι κάπως ηρωνικό που πριν από 10 χρόνια ακριβώς, τον Σεπτέμβριο του 2006, υπέβαλα και παρουσίασα σε αυτήν ακριβώ την Επιτροπή Πολιτικών ε, Ελευθεριών, Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων την αναθεώρηση και τη σχετική έκθεση που είχε εκπονηθεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεμελιώδη Δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη τη χρονιά. Θα θυμάστε ότι η ομάδα αυτή ε, ιδρύθηκε το 2002 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν ετοίματο του Ευρωκοινοβουλίου γιατί Είσαστε τότε πεπισμένοι ότι έπρεπε να δημιουργήσει ένα τέτοιο δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, ώστε να ενώσουν τις γνώσεις των ανεξάρτητων νομικών και να εκπονούν ετησίω έκθεση για τα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, και μάλιστα σε βάση συστηματική. Η μελέτη στην οποία αναφερθήκατε και η οποία μοιράζεται στην αίθουσα που ζητήθηκε από την ε, Ομάδα για τα Συνταγματικά και Θεμελιώδη Δικαιώματα μετά από έντοιμα της Επιτροπής ΛΥΠΕ δείχνει το γενικό αρχιτεκτόνημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της προστασίας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασιστήκαμε στο έργο του δικτύου των ανεξάρτητων εμπειρογνωμών μεταξύ 2002 και 2007, αλλά και την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη 15 Οκτωβρίου 2003 για τι αξίε, τι θεμελιώδει αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μελέτη μα κυρίω προτείνει να ζητηθεί από τον ΦΡΑ, τον Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, ε, και να ζητάτε ετησίω μια έκθεση που να καλύπτει, να καλύπτει όχι μόνο το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το δίκαιο που αφορά την, ε, το σεβασμό του, αλλά την κατάσταση όλων των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου στην ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό θα επέτρεπε στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο να εκπληρώσουν τα καθήκοντά του βάσει του άρθρου 7 για τη, λειτουργία, τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να επιδιώκουν ε, διαρκώ τον ώστε να διασφαλιστεί η συνεκτική, αντικειμενική και αμερόληπτη μη επιλεκτική αξιολόγηση της κατάστασης των 100 μελών. Έτσι, η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να γίνει πιο δυναμική και όχι απλώ ε, να αντιδρά στι καταστάσει με ε, εξουσίε που να βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη θέσπιση τη εσωτερική αγορά ε, επίση στον τομέα των ελευθεριών, τη ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Υπάρχει μια μετατόπιση λοιπόν, μετατόπιση προ αυτό που ονομάζουμε κύκλο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μια τέτοια πορεία θα εξασφάλιζε περισσότερη εξοπιστία και συμμόρφωση με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΙΕ. Πολλοί είναι οι φορεί σήμερα που ζητούν περισσότερε σχέσει συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Ήδη τον Μάιο του 2014 το Συμβούλιο τη Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση επανεπιβεβαίωσαν την διαρκή του δέσμευση να εμβαθύνουν τι σχέσει συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Συμβουλίου τη Ευρώπη στου φορεί ε, του συμβουλευτικού και τη παρακολούθηση μεταξύ του Συμβουλίου τη Ευρώπη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να συγκλίνουν τα πρότυπα του πρώτου και τη νομοθεσία τη δεύτερη και βάσει του Μνημονίου Κατανόηση του 2007. Οι μηχανισμοί ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι πολύ σκόπιμοι στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εκεί η ανάγκη για σχέση συνεργασία είναι προφανές, ε, προφανής. Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσει σήμερα ένα ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα μπορούσε να είναι το σημείο αφετηρίας για να προχωρήσουμε σε μια αναθεώρηση της χάρτας των κοινωνικών δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης που είναι μέρος του κοινοτικού κεκτημένου έτσι κι ή πάντων έχει γίνει δεκτό από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα θεμελιώδη και κοινωνικά δικαιώματα πρέπει να γίνονται αντιληπτά ω θεμελιώδη δικαιώματα που είναι γενικέ αρχέ που διέπουν το ευρωπαϊκό δίκαιο πέραν και πάνω από τα κοινωνικά δικαιώματα που τόσο άλλο συμπεριλαμβάνονται στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οι διατάξει αυτέ τη αναθεωρημένη κοινωνική χάρτα θα μπορούσαν με τη σειρά του να λάβουν υπόψη τα πορίσματα τη ε, Επιτροπή για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του ΟΗΕ, καθώ και τι αποφάσει που εγκρίνονται από το φορέα αυτό. Θα μπορούσε η ε, δράση αυτή να αξιοποιήσει και την παρακολούθηση από φορεί του Συμβουλίου τη Ευρώπη και από άλλου φορεί ανά τα κάτι μελη που είναι υπεύθυνα με την παρακολούθηση τη υλοποίηση τη άσκηση των Θεμελιώδη δικαιωμάτων, ώστε η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να βασίζονται σε μια ανδιαφυσβήτητη πηγή πληροφοριών και να ε, συμμορφούνται πλήρως με τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 2 τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αντί να αποδυναμώνεται ο ρόλος των φορέων λοιπόν του Συμβουλίου της Ευρώπης, ίσα ίσα έτσι θα ενισχυόταν η εγκυρότητα των πορισμάτων τους, και αυτά τα πορίσματα θα εντάσσονταν στις διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, επίσης όλη η διαδικασία χαράξης νομοθεσίας και πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας επιλογής θα επέτρεπαν την ευκολότερη σύγκριση για το πώ έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν πολύ χρήσιμο αυτό για να επιτρέψει την ε, δυναμική χάραξη πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι μόνο να αντιδρούμε σε παραβιάσει όπω συχνά συμβαίνει και να εντοπίζουμε ποιε αρμοδιότητε αναλογούν στην Ένωση και ποιε μπορούν να ασκηθούν ή σε ποιε μπορεί να αναποτεθεί, να αναποτεθεί η εμπιστοσύνη τη, ώστε να υπάρξει ε, τέτοιο κλίμα εμπιστοσύνη μεταξύ Ένωση και κρατών μελών. Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Στην ανακοίνωση τη 15η Οκτωβρίου 2003 και βάσει του έργου του Δικτύου των Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή θεώρησε ότι ε, θα πρέπει να μπορεί το έργο του Δικτύου να, να εντοπίζονται οι ανομαλίες και οι παρατυπίε στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όταν αυτές οι παραβιάσεις εμπίπτουν εντός του πεδίου του άρθρου 7 τη ε, Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε λοιπόν το δίκτυο να προτείνει λύσεις, να προτείνει άσκηση ένδικων μέσων για να διορθωθούν οι παραβιάσεις, και η παρακολούθηση θα έπρεπε να έχει περισσότερο προληπτικό ρόλο, ώστε να δίνει ιδέες για να επιτύχουμε τον κοινό χώρο ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας, καθώς και να εντοπίζει τάσεις ε, που προσωμιάζουν μεταξύ των μελών, ώστε να ε, διέπονται από τις ίδιες γενικές αρχές όλες οι πολιτικές η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τα υπόλοιπα θεμελιώδη δικαιώματα όπως προβλέπονται από την ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται σαν να προβλέπουν ε, περιορισμούς και φραγμούς. Όμως θα μπορούσε να είναι ε, μία πηξίδα που να κατευθύνει τη δράση μας ε, και να δίνει δυνατότητε. Δεν έχει συγκεκριμένη πολιτική θεμελιωδών δικαιωμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αναδειχθεί μια τέτοια πολιτική θα πρέπει τα θεμελιώδη δικαιώματα να φανούν όχι μόνο ένα παράγοντα περιοριστικό, αλλά πηγή έμπνευση για νομοθετικέ πρωτοβουλίε, για χάραξη πολιτικών, για διαθεσμικό διάλογο, αλλά και για διαπραγματεύσει μεταξύ των 100 μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Συμβουλίου. Η προετοιμασία από τον ΦΡΑ μια ετήσια έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του κράτου Δικαίου και τη Δημοκρατία στην Ένωση θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο σημείο αφετηρία, ένα εφαλτήριο, ώστε να ε, αρκεί μάλλον να οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο χάραξη πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, βάσει του άρθρου 7 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαν να οργανώνουν συζήτηση ε, βάσει τη έκθεση αυτή του ΦΡΑ και επίσης αυτή να καθοδηγεί την Επιτροπή στον να εντοπίζει τις πρωτοβουλίε που θα πρέπει να προτείνει βάσει των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τις συνθήκες ω προ την νομοθετική πρωτοβουλία και την ανάληψή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ίδια την Επιτροπή. Επίση, μια τέτοια έκθεση θα μπορούσε να συνδυάσει την νομική ε, μελέτη με την ανάλυση των ε, πολιτικών αναγκών, κυκλικών πολιτικών αναγκών ε, για τα θέματα αυτά. Θα μπορούσε λοιπόν να χρησιμοποιείται ένα σύνολο δικτών για να μετράτε συγκεκριμένα η πρόοδο στη βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου, αυτό που ονομάζονται διαρθρωτικοί δείκτε, αλλά και στη χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών που σκοπό την πλήρη πλήρη άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αυτό που ονομάζουμε ενδράση δείκτε, αλλά και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί. Ε, δείκτε επί των αποτελεσμάτων. Τέλο, ο οργανισμό έχει αναπτύξει μια σειρά από μεθόδου τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων ποσοτικέ μελέτε, ποιοτικέ μελέτε, συνεντεύξει, ομαδικέ συνεντεύξει, ε, παρακολούθηση τη ε, έκφραση των μέσων μαζική ενημέρωση, όχι μόνο στο νομικό πεδίο, αλλά για να δει και τι συμβαίνει στην πράξη και ποια είναι η αντίληψη για τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από του πολίτε. Έτσι, ο ΦΡΑ θα μπορούσε να συμπληρώνει όσα κάνουν οι υπόλοιποι που παρακολουθούν το πλαίσιο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλα αυτά ω πορίσματα να υποβάλλονται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν υποτιμώ ούτε στιγμή τι δυσκολίε μια τέτοια προσπάθεια και τι αλλαγέ που θα απαιτήσει. Η Επιτροπή το Κοινοβούλιο, ο Οργανισμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, εκπονούν ξεχωριστές εκθέσεις στα πλαίσια του ετήσιου διαλόγου του Συμβουλίου για το κάτω δικαίου. Θα είχαμε ένα και μόνο πολιτικό κύκλο που να βασίζεται σε πληροφορίε, οι οποίες αντικειμενικώ και αμεροληπτω θα συλλέγονται ε, από όλα τα κάτι μέλη. Θα υπάρχουν προβλήματα βεβαίω. Υπάρχει το πρόβλημα τη νομική βάση Υπάρχει το πρόβλημα που πώς να συσχετίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, έννοιες που είναι κάπως ασαφές πώς μπορούμε να συνδυάσουμε, αλλά διαρκώς ε, βελτιώνεται η κατανόησή τους και η αποσαφήνισή τους, ε, κυρίως χάρη στην Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου, για να προχωρήσουμε προς αυτό το κύκλο χαράξης πολιτικής. Η θέση που λαμβάνει η μελέτη, και θα κλείσω με αυτό, είναι ότι οι ανησυχίε που έχουν ακουστεί τα τελευταία χρόνια για τι εξελίξει του κράτου δικαίου στην Ουγγαρία και την Πολωνία, η κατάργηση τη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και η διαχείριση τη λεγόμενη κρίση των προσφύγων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα μέσα του 2015, η αποτυχία να επιτελέσουν σημαντική πρόοδο λόγω χάρη για, την, για το θεματολόγιο τη μη διακριτική μεταχείριση στην Ένωση, την ε, συμπερίληψη των, ανθρωπίνων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην οικονομική διακυβέρνηση, τα δικαιώματα του παιδιού, Όλα αυτά είναι συμπτώματα ενός βαθύτερου προβλήματος της ανικανότητας της Ένωσης να βρει εφάνταστες λύσεις για τις διάφορες μορφές κρίσης που αντιμετωπίζει και να αναθεωρήσει τις αξίες της. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει εδώ να, καθορι... ένα καθοριστικό ρόλο, ε, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να σεβαστεί τις υποσχέσεις της και δημιουργώντας μια εσωτερική αγορά που να συνδυάζει επίσης ένα κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Μια ένωση δικαιωμάτων. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, το λόγο έχουν οι ευρωβουλευτές που θέλουν να παρέμβουν. Ο κύριος Νάγκη ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τόσα είπατε, για τα μηνύματα που μας μεταφέρατε. Δύο σημεία θέλω να θίξω. Πρώτον, θέλω να υπογραμμίσω το ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ήμουν μέλο στο Συμβούλιο της Ευρώπης πριν και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τη σημασία που έχει το σώμα αυτό, ο οργανισμός αυτός, προκειμένου να προωθηθούν όλες οι συστάσεις και όλα τα ψηφίσματα τα οποία έχουν ξεκινήσει από εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει το δρόμο και να βοηθήσει τις χώρες που είναι μέλη στο Συμβούλιο της Ευρώπης και δεν είναι μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, θέλω να αντιδράσω στο μήνυμα του Επιτρόπου Τίμερμανς. Ναι, συμφωνώ, υπάρχουν φόβοι Υπάρχουν οι πραγματικές απειλές και υπάρχουν και οι εικονικές απειλές. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε στο κοινό, στον κόσμο, στους πολίτες, ότι είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε στις πραγματικές απειλές. Θα ήθελα επίσης να πω ότι πρέπει να διαλύσουμε τις απειλές, είτε είναι μεγάλες είτε μικρές. Μπορεί να ακούγεται λαϊκίστικο. Μιλάμε για τις απειλές στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, αλλά πρέπει να παίρνουμε υπόψη μας και τις πιο μικρές απειλές και να τις διαλύουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα στη σειρά ο κύριος Σόγκορ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θυμάμαι στην έκθεση ΦΡΑ την προηγούμενη φορά είχαμε αναφερθεί στα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες, τους ΛΟΑΔΑ και τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες. Στην έκθεση της Επιτροπής βλέπω μια πολύ μικρή μνήα για τον πολιτιστικό και γλωσσικό διάλογο. Η έκθεση ΦΡΑ τουλάχιστον λέει ότι τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι υπάρχει διάκριση σε βάρος εθνικών μειοτήτων. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των μεταναστών και των ε, μειονοτήτων βάσει της σεξουαλικής προτίμησης. Πώς μπορούμε να συλλέξουμε στοιχεία, γιατί δεν έχουμε στοιχεία, αν κάποιες χώρες αρνούνται την ίδια την ύπαρξη τέτοιων μειονοτήτων. Και δεν μιλάω και για τις χώρες που έχουν νόμους κατά τέτοιων μειονοτήτων ή τιμωρούν τους πολίτες τους οι οποίοι χρησιμοποιούν τη δικιά τους γλώσσα. Ή όταν προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τη, δική, τη διπλή γραφή. Τι γίνεται, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ελφανία κλπ. Δεν τα ξέρετε εσείς τι συμβαίνει. Να σας τα πω εγώ. Δεν έχω τώρα χρόνο να μπω σε λεπτομέρειες και ούτε θέλω. Αλλά αν θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά αυτά που είπατε, για παράδειγμα για τον νέο μηχανισμό, τον περιμένω. Και ελπίζω ο νέος αυτός μηχανισμός να πάρει περισσότερο στα σοβαρά αυτά τα προβλήματα του 40 εκατομμύρια ανθρώπους που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και οι χώρες όπου ζουν δεν τους παίρνουν υπόψη σοβαρά. για να το πω ευγενικά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν μερικές χώρες δεν θέλουν καν να σκεφτούν ότι υποσχέθηκαν ότι θα τηρήσουν τα κριτήρια της Κοπεχάγης και άρα κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα και απέναντι στις εθνικές μειονότητες προφανώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το γεγονός ότι ο κύριος Τίμερμανς δεν είναι εδώ σήμερα σε αυτή τη συνεδρίαση, για μένα είναι ε, ενδεικτικό της κατάστασης της δημόσιας συζήτησης για το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και ο κύριος Τίμερμανς επιλέγει ε, να μην ε, ασκεί την ευθύνη που έχει ε, ως εκπρόσωπος ενός θεσμικού οργάνου, ε, θα πρέπει στην ουσία να μας δικαιολογήσει γιατί το κάνει. Εκτός αν θεωρεί ότι είμαστε διακοσμητικό σώμα και ότι δεν έχουμε ουσία. Η δήλωση που δόθηκε εκ μέρους του, που διαβάστηκε χείρε εδώ, δεν ε, περιλαμβάνει λεπτομέρειες, αλλά λέξεις δυνατές και ηχηρές όπως ε, μίσος ε, και φόβος. Είναι μια ρητορική μίσους ίσως, αν όχι είναι ρητορική αποκλεισμού από τη δημόσια συζήτηση και με αυτόν τον τρόπο αρνείται να κάνει σοβαρή συζήτηση για τη μετανάστευση. Κάθε φορά που μιλάμε για την μυσαλλοδοξία στην πράξη, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη σιωπή, ακόμα και στις περιπτώσεις που οι συνθήκες το απαιτούν. Εμείς ε, όλο και λιγότερες πληροφορίες ε, παίρνουμε. Όλο και περισσότερες πληροφορίες παίρνουμε για διωγμούς χριστιανών, για μίσος κατά των χριστιανών, για διωγμούς ε, χριστιανών στα κέντρα των προσφύγων και των μεταναστών. Υπάρχουν και σχέδια ψηφίσματος στο Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Να πω ότι το Γερμανικό Συμβούλιο μας έχει των Ανατολικών Εκκλησιών μας έχει ενημερώσει ότι ε, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και δεν υπάρχουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Και αν, όπως είπε και ο κύριος Σόγκορ πριν από λίγο, αν το σώμα που εκπροσωπεί ταυτόχρονα δύο μορφές μειονοτήτων, γιατί εκπροσωπούν και τις εθνοτικές και τις θρησκευτικές μειονότητες, το Συμβούλιο δηλαδή για τις Ανατολικές Εκκλησίες, αν αυτό το σώμα λοιπόν κάνει αυτή τη δήλωση, οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υποχρεωμένες ε, να διεξαγάγουν διάλογο με ε, τις θρησκευτικέ οργανώσεις και το θρησκευτικό κόσμο, όπως εγγράφεται στις συνθήκες, θα πρέπει τουλάχιστον να επιβεβαιώσουν αυτά τα στοιχεία, να ενδιαφερθούν. Επίσης βλέπουμε ότι υπό τη σκέπη των ιδεολογικών ε, αφορισμών ε, στην ουσία ε, παραμένουμε σιωπηροί ενώπιον αυτών των θεμάτων. Δεν έχουμε ακούσει ούτε μία λέξη για το μίσος κατά των χριστιανών. Κάποιες φορές ε, ε, δεν μπορούμε καν να καταγράψουμε τα πραγματικά γεγονότα, από όλο δε μάλλον τις σκέψεις. Ε, έχω την ελπίδα ότι είχα την ελπίδα ότι αν ήταν εδώ ο κύριος Τίμερμανς θα μπορούσα να το ρωτήσω για τις παράνομες πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι έχει βάλει το όνομα της σε δράσεις που απευθύνονται κατά της χώρας μου που αμφισβητούν και οι νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Βέβαια, όχι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οπότε έτσι τις ξεπερνάμε. Είναι μια πολιτική ευθύνη, λοιπόν, η οποία δύσκολα τίθεται στην πράξη, όταν η συζήτηση στην ουσία απλώς αντιμετωπίζεται ως ανταλλαγή απόψεων δεν αντιμετωπίζεται ως επερώτηση στις αρχές που ασκούν τα καθήκοντά τους έναντι των πολιτικών ομάδων και εκπροσωπούν την επιτήρηση αυτών των δράσεων. Λυπάμαι πολύ και λυπάμαι που δεν μπορώ να μιλήσω στον κύριο Τίμερμαν σε αυτή την επιτροπή και δεν θα μπορέσω να του μιλήσω στο μέλλον, ούτε και στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Σόφη Ινφελτ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, είναι μεγάλη μου χαρά που βλέπω ε, εδώ τον κύριο Ντεσρόιτερ ξανά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Θυμάμαι ε, την έκθεση για το Concord που το, εκείνη την εποχή είχε πολύ περίεργες ε, επιπτώσεις. Άκουσα την παρουσίασή σας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα που έχουν γίνει, υπάρξει, αλλά φαίνεται ε, ότι ούτως ή άλλω η αλλω η Επιτροπή αυτή τη στιγμή συντάσσει μία έκθεση για ένα σύστημα βάσει του οποίου τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα θα τηρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Θέλω να ακούσω τα σχόλιά σας γι' αυτό. Δεύτερον, ερώτηση στον κύριο Μωρίγιο και μέσω αυτού στον κύριο Τίμερμανς. Λυπάμαι που ο κύριος Τίμερμανς δεν είναι εδώ. Ειδικά σε αυτό το πάνελ σήμερα θα ήθελα να ρωτήσω, να ζητήσω από την Προεδρία της Επιτροπής να ζητήσει από τον κύριο Τίμερμανς να έρχεται πιο συχνά σε αυτήν την Επιτροπή, γιατί στην άλλη Επιτροπή στην οποία είμαι μέλος έχουμε πάρα πολύ συχνές ανταλλαγές απόψεων με τους αντίστοιχους επιτρόπους που έρχονται σε μας κάθε τρεις μήνες ή κάτι τέτοιο. Θα ήταν πολύ χρήσιμο λοιπόν. Έχω λοιπόν κάποια ερωτήματα, γιατί βέβαια μόλις πήραμε την έκθεση και δεν είχαμε το χρόνο να τη δούμε, αλλά ακούγοντας την παρέμβασή σας και βλέποντας το, τα περιεχόμενα της έκθεσης, Και βάσει των εκθέσεων που έχουμε λάβει τα τελευταία χρόνια, θεωρώ ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ αυτού που βιώσαμε και βιώνουμε στις καθημερινές μας συζητήσεις και σε αυτό που παρουσιάζει η έκθεση. Διαβάζεις την έκθεση και όλα πάνε καλά και η Κομισιόν είναι ο προστάτης ε, και ο πρώτος που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως τελικά εμείς αμφισβητούμε ακόμα και το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα ανθρώπινα δικαιώματα στις προτάσεις της. Θεωρώ ότι δεν τα λαμβάνει πάντοτε πλήρως και επαρκώς υπόψη της. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα για προτάσεις που σχετίζονται ας πούμε με την μάχη κατά της τρομοκρατίας Επίσης θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει πλήρως υπόψη την ομολογία που, στην οποία βασίζεται η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει επίσης αξιολόγηση επιπτώσεων που να συνοδεύει τις ε, πολιτικές για την πάταξη της τρομοκρατίας. Και είναι ευαίσθητε αυτές οι πολιτικές. Γιατί λέει συνεχώς η Κομισιόν ότι δεν έχει χρόνο ε, για να δει πώς επηρεάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης υπάρχουν διάφορα κοινοβουλευτικά ερωτήματα και επιστολές που έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή για αυτά τα θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συνήθως δεν λαμβάνουμε απάντηση, ακόμα και όταν πάρουμε δεν υπάρχει μια συνέχεια, μια παρακολούθηση, δίνεται η εντύπωση ότι η Κομισιόν δεν έχει μεγάλη θέληση να το κάνει. Ένα παράδειγμα, μας ανησυχούν ιδιαίτερα οι συνεχείς προσπάθειες στη Λιθουανία να περάσει νομοθεσία κατά τον ΛΟΑΔ μέσω του νόμου κατά της προπαγάνδας που τώρα εφαρμόζεται. Πραγματικά ανησυχούμε ιδιαίτερα για το πώς εφαρμόζεται. Ακούσαμε από την Κομισιόν πριν από ένα χρόνο ότι το εξετάζουν. Και τώρα περιμένουμε τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το θεωρώ απίστευτο. Θα ήθελα επίσης να μάθω τι πρόκειται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει τις δικές της επιδόσεις ως προς την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα έπρεπε να έχει λίγο περισσότερο θάρρος, θα έλεγα. Και πραγματικά Λυπάμαι που κάθε φορά πρέπει να απευθύνω τα ερωτήματα στον καημένο τον κύριο Φωνσέκα Μωρίγιο και πάντοτε αυτός ε, να είναι ε, αντικείμενο του θυμού μου και τα δικά σας θεμελιώδη δικαιώματα παραβιάζονται. Νομίζω λοιπόν ότι ο κύριος Τίμερμαν θα έπρεπε να είναι εδώ να απαντήσει στις ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα να ακούσω την απάντησή σας. Ε, Ο κύριος Κάρσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, συχνά αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπου οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας η έλλειψη νόμων οδηγούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτός της επικρατείας μας, όπου ε, οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανοχή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων οδηγούν σε πραγματικές ε, παραβιάσεις ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη μιλήσαμε για τους ξένους μαχητές σήμερα, αλλά κάποιες φορές Έχουμε και το πρόβλημα της δράσης ευρωπαϊκών εταιρεών ή επιχειρήσεων που λειτουργούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραβιάζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και εκεί αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπου τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξάγουν στρατιωτικές υπηρεσίες, ε, ιδιωτικές μάλιστα, στο εξωτερικό. Και κάποιες φορές Αυτά συνδυάζονται με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του διεθνούς δικαίου. Και κάποιε φορές υπάρχει απουσία ανάληψης ευθυνών των ανθρώπων που δρούν κατά αυτόν τον τρόπο ή και έλλειψη λογοδοσία. Οι χώρες όπου λειτουργούν τους παρέχουν ατιμορρησία και ασυλία. Επίση οι εταιρείε αυτές πολύ συχνά είναι ε, καταγεγραμμένες στα δικά μας κράτη-μέλη που όμως δεν ενδιαφέρονται να εκδικάσουν τέτοιες υποθέσεις. Και πολλές φορές εντοπίζουμε κενά και ελλείψεις εντός της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η οδηγία περί υπηρεσιών ε, εξαιρεί τις θετοτικές υπηρεσίες και κάποιες άλλες υπηρεσίες ε, ασφαλείας. Δεν ξέρουμε γιατί. Γιατί αυτή η παρέκκληση προβλέφθηκε στη διάρκεια των ε, δραστηριοτήτων Τη χάραξη ε, τη ε, πρότασης μάλλον νομοθεσίας, ίσως λόγω των ομάδων πιέσεων, των λόμπι που το ζήτησαν. Παρ' όλα αυτά, αυτή η παρέκκληση υπάρχει. Και βεβαίως η ΕΕΔ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησαν να ε, λάβουν υπόψη τις δράσεις των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν τις υπηρεσίες ασφαλείας ή στρατιωτικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σεβαστούμε τις δικές μας αρχές και στη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλές φορές ε, τοποθετούνται με πολύ έντονες εκφράσεις, κάποιες φορές επιθετικές κιόλας, υπέρ της ε, διατήρησης του status quo και του τρόπου με τον οποίο οι εταιρείε που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πολυμερή συμφωνία του Μοντρέ είναι ε, δυστυχώς μη δεσμευτική νομικός, οπότε κάτι πρέπει να προβλέψουμε που νομικός να δεσμεύει τους πάντες. Να πω το εξής στον εισηγητή. Θα πρέπει να προσέχουμε το τι συμβαίνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι κάνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρώπη. Διότι δεν θέλουμε παραβιάσει των θεμελιωδών δικαιωμάτων από εταιρείε που έχουν την έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω αποτέλεσμα τη αδιαφορία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Σκρίπεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω ερώτηση προς τον κύριο Γκρούντεν. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Μιλήσατε για την ε, ευθυγράμμιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ε, ομιλία σας. Οι εκφράσεις μίσους είναι μία περίπτωση. Ένας χώρος πολύ προβληματικός κατά την άποψή μου διότι οι εκφράσει μίσου ενό ε, ανθρώπου καταπιέζει την ελευθερία έκφραση κάποιου άλλου. Και δημιουργείται ένα ειδικό χώρο διεπαφών εδώ. Το ε, Συμβουλίο τη Ευρώπη έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για την προστασία τη άσκηση θρησκευτικών ε, δογμάτων ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το δικαίωμα να προβάλλει κανεί αντίρρηση συνείδηση. Εδώ μπορείτε να μα πείτε τι συμβαίνει με την ανεξιθρησκεία και την ε, ελεύθερη έκφραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα γίνονται σεβαστές αυτές οι ελευθερίες χάρη στις εκθέσεις λόγου, χάρη οι χριστιανοί, κάποιες φορές οι εκκλησίες τους, τα πίμνια, μπορεί να απειλούνται λόγω της άσκησης των θρησκευτικών τους πεπιθήσεων, των πρακτικών τους ή τέλος πάντων της απλής έκφρασης των απόψεών τους. Πώς αποφασίζετε, αυτή είναι η ερώτησή μου, ότι αυτά που λέω μπορεί να διέπονται από μίσους. Πώς ασκώ την δυνατότητά μου να διαφωνήσω με την έκφραση σεξουαλικών προσανατολισμών κάποιων, λόγω χάρη. Μπορώ να διαφωνώ με τις ε, συνήθεις άλλων. Είναι δικαίωμά μου. Αν όμως βλάψω κάποιον ή διαπράξω ένα έγκλημα, δίκαιο επίσης είναι ο νόμος να με διώξει. Δεν μισώ κάποιον ο οποίο αυτοπροσδιορίζεται ω ομοφυλόφιλο, αλλά δεν ανάγκη να συμφωνώ με τι πρακτικέ που ασκεί και τι εκφράσει του. Ε, θα πρέπει λοιπόν την ελευθερία να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις να τη διατηρήσουμε, να μπορούν να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις. Καθένας που θέλει να κηρύξει την άποψή του θα μπορούσε να εκφράσει και τη διαφωνία του σε σχέση με κάποιες πρακτικές. Πρέπει να επιτρέψουμε και ένα χώρο ελευθερίας. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβλέπει νόμους για τα θέματα αυτά. Γνωρίζετε ότι η πηγή των εκφράσεων μίσους στη Ρωσία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν κατά του οποιοδήποτε στοιχείο δεν ήταν κομμουνιστικό. Έρχε, έρχομαι από μια χώρα που είναι, ήταν μέρος του Σοβιετικού μπλοκ και το έχω ζήσει αυτό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μισούμε στην κοινωνία αυτή, να δεν μπορούμε και να τιμωρούμε κάποιον για τη μισή. Ό,τι και αν λέτε, ε, σίγουρα δεν μα αρέσει ο θρησκευτικό φανατισμό, αλλά δεν μπορεί κανεί να τιμωρείται για τι απόψει αυτέ. Δεν μου αρέσει το τζιχαντιστικό Ισλάμ. Προφανώ είναι μία σέκτα. Αλλά μπορούμε να τιμωρούμε του ανθρώπου για τι απόψει του και τι πρακτικέ του έτσι απλά. Πού είναι τα όρια μεταξύ των μαχητών του Άιζη που διαπράττουν ένα έγκλημα και την έκφραση μίσου κατά τη χριστιανοσύνη, λόγου χάρη. Τα ξένα μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα λένε ότι όσοι εκφράζουν μίσος θα πρέπει να διώκονται για τις απόψεις τους. Πού είναι το όριο για την Λετωνία, όπως αναφέρθηκε και από την ε, συνάδελφο Ιντεβέλτ, η Λετωνία έχει το δικαίωμα να μην επιτρέπει τη διάδοση πρακτικών λαόδ, ΛΟΑΔ μάλλον ή των ομοφιλοφιλικών τάσεων και η Ρωσία έχει το δικαίωμα να μην επιτρέπει τις αμβλώσεις. Δεν μπορούμε να το ονομάσουμε αυτό μίσος ή έκφραση μίσους και πώς ε, φτάνουμε και σε μια υπόνοια ότι όλα αυτά θα έπρεπε ίσως να τιμωρούνται. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαριάς, τελευταίος ομιλητής. Uh, Chairman, I'm going to continue in Greek, if I may. Uh, Ευχαριστώ, θα συνεχίσω ελληνικά, αν μπορώ. Σε σχέση με την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την πλευρά της Τρόικας και του Eurogroup, διότι η Τρόικα είναι ένα όργανο το οποίο νομικά δεν υφίσταται, αλλά στην πράξη λειτουργεί αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και, την, και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Και παίρνει σημαντικές αποφάσεις όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Κύπρο. Και οι αποφάσεις αυτές, όπως και οι αποφάσεις του Eurogroup, το οποίο συνεδριάζει ω εκπρόσωπο των δανειστών, όπω και οι αποφάσει του ESM, που είναι διακρατικός διεθνής οργανισμός, αλλά παίρνει σημαντικές αποφάσεις για την χρηματοδότηση, της, ε, τον, την δανειοδότηση της Ελλάδος ή και των άλλων κρατών που ήταν σε μνημόνια. Οι αποφάσεις που παίρνουν λαμβάνονται υπό τη μορφή μνημονίου, Memorandum of Understanding. Εκεί λοιπόν σε αυτό το μνημόνιο, το οποίο επιβάλλεται στις κυβερνήσεις και το ξέρουμε, διότι αν δεν το αποδεχτούν οι κυβερνήσεις δεν πρόκειται να πάρουν χρήματα, και το οποίο συντάσσεται από την Τρόικα και αποστέλλεται στις κυβερνήσεις για υπογραφή, εκεί λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα κράτη. Και οι δεσμεύσεις αυτές προκαλούν συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα το οποίο παραβιάζει πολύ συγκεκριμένα δικαιώματα. Παράδειγμα, υπάρχουν μέτρα τα οποία αφορούν την μείωση των συντάξεων. Η σύνταξη όμως είναι ατομικό δικαίωμα και μάλιστα δικαίωμα ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται και προστατεύεται από το άρθρο 17. Όταν σου μειώνουν τη σύνταξη όπως μειώθηκαν στην Ελλάδα κατά 40% σου περιορίζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Όταν σου μειώνουν τη σύνταξη παραβιάζεται το άρθρο 25 που είναι το δικαίωμα των ηλικιωμένων στην αξιοπρεπή διαβίωση. Όταν σου μειώσουν τις, ε, τους μισθούς παραβιάζεται παραβιάζονται πολλά συγκεκριμένα δικαιώματα σε σχέση με την διαβίωση των προσώπων. Επίσης, το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Όταν μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες και δεν έχεις καλή εκπαίδευση, παραβιάζει το άρθρο 14. Όταν α, ε, σου πάρουν μέτρα τα οποία δημιουργούν προβλήματα και μειώνουν την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, παραβιάζει το άρθρο 36, που είναι η παραβίαση σε υπηρεσίες γενικών οικονομικών συμφερόντων. Όταν παίρνονται μέτρα για την περίθαλψη και τα νοσοκομεία παραβιάζεται το άρθρο 35. Όταν μειών, αλλάζει το συνταξιοδοτικό όπως έγινε στην Ελλάδα παραβιάζεται το άρθρο 34. Τι θέλω να πω. Ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια γκρίζα ζώνη. Ποιο είναι αυτό που θα ελέγξει την παραβίαση δικαιωμάτων από πλευρά Τρόικα. Διότι εν προκειμένου η Κομισιόν δεν ενεργεί ω Κομισιόν, γιατί δεν έχει καν δικαίωμα η Κομισιόν να μιλήσει για θέματα κοινωνική ασφάλιση. Αυτά δεν ανήκουν στι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει καν δικαίωμα να μιλήσει για τον ελάχιστο μισθό, διότι αυτό υποτίθεται ότι ανήκει στα κράτη-μέλη. Κι όμω παρεμβαίνει. Το ίδιο κάνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ίδιο κάνει και το Eurogroup. Και όλα αυτά παράγουν πλέον ένα δίκαιο το οποίο επιβάλλεται επί των πολιτών και ταυτόχρονα παραβιάζει τα δικαιώματά τους. Πού θα προσφύγουν οι πολίτε οι οποίοι θέλουν να το κάνουν. Έχω κάνει αυτό το θέμα, το έχω πει επανειλημμένα και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Επιτροπή Αναφορών. Και έρχεται η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας, η κυβέρνηση της Κύπρου και νομοθετούν και παίρνουν μέτρα. Και έχουμε θέσει ερώτημα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη δράση των κρατών. Και εκεί μας απήντησε η Κομισιόν ότι ξέρετε κάτι, αυτές δεν είναι δράσεις που έχουν σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά είναι δράσεις που έχουν σχέση με τα κράτη. Λες και δεν είναι η Κομισιόν ή δεν είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που επιβάλλει τους όρους για τα NPL σφερπίν και για τις εξώσεις αυτή τη στιγμή που γίνονται στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν το σημαντικό θέμα το θέτω όχι μόνο I'm going to finish in seconds. Ε, αυτό το σημαντικό θέμα λοιπόν το θέτω όχι μόνο σαν βουλευτή αλλά και σαν πανεπιστημιακό. Γιατί διδάσκω, είμαι καθηγητή θεσμών Ευρωπαϊκή Ένωση στο Πανεπιστήμιο τη Κρήτη. Δεν μπορεί να έχουμε γκρίζε ζώνε σε αυτό το θέμα. Και είναι κάτι που δεν το αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το έχουμε θέσει σε ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ορισμένε φορέ το θίγει. Πρέπει λοιπόν και αυτή την πλευρά να δούμε πώ θα την αντιμετωπίσουμε. Διότι έτσι διαμορφώνεται ένα κλάδο δικαίου που είναι μια γκρίζα ζώνη που περιορίζει τα δικαιώματα τα θεμελιώδη και όμως δεν μπορεί κανείς να ελέγξει την νομιμότητα. Αυτά λοιπόν πρέπει να μας προβληματίσουν έντονα, ιδίως για την Ελλάδα, όπου αυτή τη στιγμή γίνεται μια μαζικότατη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σας ανέφερα παραδείγματα λόγω και του τρίτου μνημονίου που εφαρμόζεται. Θα πείτε να μην εφαρμόσει την νομοθεσία ελληνική κυβέρνηση. Θα σας πω, μα δεν θα της δώσουν χρήματα και νέα δανειοδότηση και δεν θα μπορεί να πληρώσει ποιον. Τον κύριο Ντράγκη. Γιατί τα ομόλογα του κυρίου Ντράγκη πληρώνουμε και τη ΕΚΟΥΤΟΥ με τα δανεικά που μα δίνουν. Το 75% των δανεικών πηγαίνει πίσω στου δανειστέ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, thank Ευχαριστούμε. Σόφιν Χετφέλτ ήθελε να παρέμβει. Ένα λεπτό όμως παρακαλώ. Ε. Ναι, ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ειλικρινά δεν μπορώ να σιωπήσω μετά τις παρεμβάσεις Γιούρε και Σχρίκερ. Βεβαίω και έχετε δικαίωμα να λέτε ότι σκέφτεστε, βεβαίω έχετε δικαίωμα στη γνώμη σα, αλλά υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο να υποστηρίζει κανεί την άποψή του ή να έχει ρητορική μίσου ή μονίμω να δηλώνει κατά τον ΛΟΑΔΑ, κάτι το οποίο δημιουργεί ένα κλίμα μέσα στο οποίο ο κόσμος δεν αισθάνεται άνετα. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε κάποιες αξίες. Μετά από αυτά που έγιναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που 50 άτομα σφαγιάστηκαν με τρομερό τρόπο, απλώς και μόνο επειδή ήταν αυτοί που ήταν, πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά τι αξίες διαδίδουμε. Θλίβαμε Οργίζομαι που ακούω αυτή τη ρητορική, την ομοφοβική, ξανά και ξανά και ξανά εδώ σε αυτό το σώμα. Και γι' αυτό ήθελα να το εκφράσω. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, δεν θέλω να αρχίσουμε μια νέα συζήτηση πάνω σε αυτό, παρακαλώ. Θα έχουμε ένα επόμενο πάνελ σε λίγο. 30 δευτερόλεπτα κι εσείς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Έχω δικαίωμα να αντιδράσω γιατί αναφερθήκατε σε μένα πριν. Κοιτάξτε, δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα. Ε, κάποιες χώρες μέλη θέλουν να υποστηρίξουν την οικογένεια σαν μια κοινωνική προδιαγραφή. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την οικογένεια ή επίσης θέλουμε να αντιδράσουμε στο Ισλάμ που υποστηρίζει την πολυγαμία ή διαφορετικές σχέσεις ανάμεσα στη γυναίκα και τον άντρα. Πρέπει να μπορούμε να το υποστηρίξουμε αυτό. Να υποστηρίξουμε την μονογαμία σε αντίθεση με άλλες κοινωνίες που δεν την υποστηρίζουν. Υπάρχουν οικουμενικές προδιαγραφές που πρέπει να γίνουν κατανοητές. Εμείς υποστηρίζουμε τη και θα συνεχίζουμε να το κάνουμε. Είναι μια χώρα μειονότητα. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε και αυτές τις μειονότητε. Ευχαριστώ. πρόεδρο. θα συζητήσουμε σε λίγο για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Αυτή είναι η σωστή πλατφόρμα για να θέσετε τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω εγώ να βγάλω συμπεράσματα, αλλά να αναφέρω το εξή. Ίσως θα ήταν καλό να καλέσουμε προσωπικά τον κύριο Τίμερμανς εδώ να έρθει να συζητήσει με την Επιτροπή μας στη Λίμπερ. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το συμπέρασμα της συζήτησης αυτής. Τώρα, θα ήθελα να δώσω το λόγο Δύο λεπτά ο καθένας παρακαλώ στους ομιλητές μας, τους εισηγητές. Ο κύριος Φονσέκα πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και για να απαντήσω όσον αφορά την γλωσσική ποικιλομορφία θα απαντήσω στα γαλλικά. Ακριβώς για να υπάρχει αυτή η πολυμορφία. Λοιπόν, θα μεταφέρω στον κύριο Τίμερμανς τα όσα άκουσα εδώ και την ε, απογοήτευσή σας που δεν ήταν εδώ σήμερα. Θα του το πω μόλις επιστρέψω στο γραφείο μου. Δεύτερον, για τις ερωτήσεις που μου θέσατε. Λυπάμαι που βρήκατε ότι η γλωσσική πολυμορφία ε, παίρνει ένα πολύ μικρό μέρος στην έκθεση. Εμείς σκεφτήκαμε ότι έπρεπε να υπογραμμίσουμε άλλα πράγματα πιο σημαντικά μέσα στο πολιτικό πλαίσιο που βρισκόμαστε σήμερα στην Ευρώπη. Αυτή είναι η μόνη απάντηση που μπορώ να σας δώσω. Όσον αφορά τώρα το θέμα των χριστιανών και το διάλογο των ε, θρησκειών. Στα τέλη αυτού του μήνα θα έχουμε την επίσημη συνάντησή μας του κ. Τίμερμαν με τις θρησκευτικέ και λαϊκές κοινότητε. Θα μεταφέρω τις θέσεις σας. Εξάλλου θα είμαι εκεί. Η Επιτροπή πρέπει να ξέρετε ότι παίρνει πάρα πολύ στα σοβαρά το άρθρο 17 και τον διάλογο με τις θρησκευτικέ και μη θρησκευτικέ κοινότητες. Για την Σοφίνη Φελτ. Μην ανησυχείτε, δεν μου επιτίθεστε καθόλου. με απρόκληση μου βάζετε και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Συγγνώμη, αν δεν ήμουν ξεκάθαρος. Η συζήτηση όμως είναι πολιτική. Εγώ εδώ μεταφέρω το αίσθημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τα όσα έγιναν στο Ορλάντο. Αγανακτούμε και αυτή την άποψη εκφράζουμε. Κατά τα άλλα τα θέματα της διαφοράς, ε, της μοφές της οικογένειας κτλ. δεν θέλω να μπω στις δικές σας πολιτικές συζητήσεις. Ξέρω ότι δεν συμφωνούμε και το άρθρο 16 για τα δεδομένα θα προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε όσο μπορούμε καλύτερα για το ΣΥΣ. Εξακολουθούμε να συζητάμε ακόμα και σήμερα με τους Αμερικανούς και αυτήν ακριβώς τη στιγμή γίνονται συζητήσεις σκληρές και δύσκολες. Τώρα για τη Λιθουανία. Παρακολουθώ από κοντά την κατάσταση στη Λιθουανία και όχι μόνο αυτό, εργαζόμαστε και σκληρά προκειμένου να πετύχουμε μια ισορροπία και να μην υπάρχει διάκριση βάσει των συνθήκων. Δεν είναι κάτι που έχουμε ξεχάσει. Τα θέματα δικαιοσύνης ε, απέναντι στους καταναλωτές επίσης προχωρούν και θα συνεχίσω και εγώ να κάνω ό,τι μπορώ. Νομίζω ότι απάντησα λίγο πολύ σε όλες τις ερωτήσεις. Τι μένει. Κατά πόσο σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα προγράμματα λιτότητας. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα και πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Αν μη τι άλλο, και στην περίπτωση της Πορτογαλίας πήγαμε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και καταλήξαμε ότι είναι αναλογικά τα μέτρα τα οποία υιοθετήθηκαν σε σχέση με το θέμα που είχε προκύψει στην Πορτογαλία. Αυτή ήταν η απόφαση του δικαστηρίου. όχι όμως στην Ελλάδα. 40% του πληθυσμού ζει υπό την ένδια και έχουμε 1,5 εκατομμύρια άνεργους. Παρόλο που η Ελλάδα πήρε 240 δισεκατομμύρια δάνειο. Πού πήγαν τα χρήματα αυτά. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα Marshall που θα μπορούσε να έχει βοηθήσει την ελληνική οικονομία και να μην είχαμε ανεργία σήμερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Παρακαλώ εσείς. Ευχαριστώ. Επειδή με ρωτήσατε κάτι, εμένα, ε, προσωπικά θέλω να απαντήσω στον κύριο Σκρίπλερ όσον αφορά τις προοπτικές για την ελευθερία έκφρασης και πώς παραβιάζονται. Η απάντησή μου είναι όχι. Φυσικά και έχετε δικαίωμα να ασκήσετε την ελευθερία σας θρησκείας, έκφρασης, ελευθερία έκφρασης βάσει του άρθρου 10. Το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι και η μόνη η οποία αναφέρεται στην υπευθυνότητα με την οποία ασκείται το δικαίωμα αυτό. Η δικαιότητα δυνατότητες να περιοριστεί αυτό το δικαίωμα αναφέρεται στην ίδια τη σύμβαση. Και πώς γίνεται αυτό. Αποφασίζεται βάσει πολύ συγκεκριμένων και περιοριστικών κριτηρίων. Κύρια, ανάλογα με το τι είναι δίκαιο και αναλογικό σε μια δημοκρατική κοινωνία. Φυσικά και μπορείτε να εκφραστείτε ελεύθερα, να πείτε πράγματα τα οποία προσβάλλουν ή ενοχλούν, αλλά υπάρχει ένα όριο. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει θέσει αυτό το όριο και οι αρχές μας, των χωρών μελών ε, δηλαδή, μπορούν και πρέπει να παρεμβαίνουν. Υπάρχει ένα όριο στην ελευθερία έκφρασης. Και επιτρέψτε μου και κάπως πιο προσωπικά να σας πω και κάτι ακόμα. Προσωπικά πιστεύω ότι νομικές κυρώσεις και ποινικέ είναι μέρος της απάντησης, αλλά θα έπρεπε να περιορίζονται πάρα πολύ και να εφαρμόζονται μόνο σε πάρα πολύ σοβαρές περιπτώσεις. Το θέμα της ρητορικής μίσους σε μια κοινωνία είναι το κατά πόσο έχουμε απάντηση σε τέτοια ρητορική που αρνείται το δικαίωμα άλλων, που επιτίθεται στην αξιοπρέπεια του άλλου. Και είναι ευθύνη μας εμάς των πολιτικών σε περίπτωση τέτοιας ρητορική μίσους να αντιδράσουμε. Αυτό θα κάνει τη διαφορά, να τοποθετηθούμε κατά μια τέτοια ρητορική και όχι να την δεχόμαστε. Αλλά αυτό είναι πιο προσωπικό. Και εγώ έρχομαι από μια τέτοια κομμουνιστική χώρα. Αυτά είχα να πω, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Um, and it's Ευχαριστώ. Είναι όντως μεγάλη χαρά που σας βλέπω, Σοφή Φέλτ. Ε, πραγματικά θαυμάζω την μνήμη σας. Οι προτάσεις που έχουν συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ενισχύσουν την παρακολούθηση των αξιών επί των οποίων έχει οικοδομηθεί η Ένωση και η μελέτη σε κάποιο βαθμό στην οποία έχει συμβάλει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και αυτή η συνεχή συζήτηση έχουν να κάνουν με τα εξή. Πρώτον, πώς τα θεμελιωδή δικαιώματα θα ενσωματωθούν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και στα μέτρα που επιβάλλονται σε χώρες ε, που έχουν κάποιο δάνειο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Αυτή είναι αυτό είναι ο πρώτος τομέας. Υπάρχει μια πρόταση από την Μπάρμπαρα Σπινέλη που μιλά για το ρόλο των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις μεθόδους εργασίας ε, των θεσμικών οργάνων. Επίσης, ποιος είναι ο ρόλος ε, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ανοιχτό ερώτημα. Τρίτο, ποιος είναι ο ρόλος των κοινωνικών δικαιωμάτων πέρα από αυτά που είναι ενσωματωμένα στο χάρτη διότι αυτή είναι μια προσωρινή και εν μέρη κωδικοποίηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε καμία περίπτωση δεν ε, αντικατοπτρίζει το κεκτημένο για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέταρτον, στο μέλλον θα προχωρήσουμε προς μια πολιτική θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, όπου οι εκθέσεις ε, δεν θα κοιτούν απλά πίσω και θα αντιδρούν ε, στα θέματα, αλλά θα προτείνουν και θα ενεργοποιούν πολιτικές. Και τέλος, μια παρατήρηση μετά από τις παρεμβάσεις σας, να πω ότι ε, στις σελίδες 21-24 της μελέτης που έχει παρουσιαστεί στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και είναι διαθέσιμη εδώ, Να αλλάξω λίγο τώρα ιδιότητα και να πω ότι ε, μιλήσω ως μέλος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να πω λοιπόν ότι αυτό που έχει συνέβη στην Ελλάδα είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό για μένα ως υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, πριν από μερικούς μήνες είχε έρθει σε εμά η ελληνική κυβέρνηση και πραγματικά αυτό που αποτιμήσαμε ήταν ε, ανατριχιαστικό. Δεν υπήρξε καμία τήρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων στην υιοθέτηση αυτών των μέτρων. Και αυτό δημιουργεί θέμα αξιοπιστία για τους παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τις τόσο ενδιαφέρουσες ε, συνεισφορές σας σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους. Και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στο άλλο πάνελ. Σας ευχαριστώ ξανά. Ευχαριστώ να προσκαλέσω στο Προεδρείο την κυρία Τόφμαν Χοϊ, τον κύριο Γκάτας, την κυρία, τον την κυρία Μελόη, τον κύριο Ιβάνοφ, τον κύριο Γκάτα, τον κύριο Κλάρκ και την κυρία Καζαρτσκίνη. Now we will start to proceed with our να ξεκινήσουμε με το δεύτερο πάνελ. Ο τίτλος είναι τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των Ρωμά, των διαφυλικών και των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Θα προσκαλέσω τους καινούριου μας ομιλητές, Πρώτος, ο Βόκτορ Μαλόι. Ή, κυρία Μαλόι διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα θέματα μειονοτήτων. Η κυρία Μαλόη είναι πολιτική επιστήμων με δίκευση στα πολιτικά και νομικά θέματα για τις εθνοτικές και εθνικές μειονότητες, τα δικαιώματά τους στο, διεθνή, στο διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς σχέσεις, ιδίως στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Επιπλέον, εκτός από διευθύντρια του ECMI, η κυρία Μαλόη είναι επικεφαλής του κλάστερ για την έρευνα, της ομάδας δηλαδή για την έρευνα, για τους πολίτες και τη διοντολογία. Κυρία Μαλόη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τις μειονότητες, επικεντρωνόμαστε στην Ευρώπη γενικώ στις εθνικές ε, μειονότητες που περιλαμβάνουν ε, ομάδες οι οποίες ιστορικά κατοικούσαν στην ίδια περιοχή για αιώνες, ε, εθνικές, ε, γλωσσικές ομάδες αλλά και Ρώμα. Σε πολλές χώρες οι θρησκευτικέ ομάδες περιλαμβάνονται επίσης σε αυτή την κατηγορία, όπως επίσης και διάφορες φυλές. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και άλλοι κανονισμοί για τις μειονότητες δεν προβλέπουν ουσιαστικά δικαιώματα για άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες προκειμένου να τους προστατεύουν και την, τον πολιτισμό τους και την ταυτότητά τους. Τα κριτήρια της Κοπεχάγης θυμίζω ότι αναφέρει διάφορα δικαιώματα αλλά δεν είδαμε να χρησιμοποιούνται πάντα. Έτσι λοιπόν, σε επίπεδο πέρα από το κράτος δεν υπάρχουν ε, διατάξεις και θετικά μέτρα για να προστατεύονται τα άτομα αυτά από την αφομοίωση για παράδειγμα. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά από σε παρακολουθεί τα πράγματα και δεν αντιμετωπίζει τα θέματα τέτοιων διακρίσεων. Τα έχει αφήσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Σύμβαση για την Προστασία των Εθνικών Μειοντήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης πάντα. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει γιατί πρώτα απ' όλα πολλές χώρες δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση πλαίσιο, αλλά επειδή και η προστασία αυτή δεν προβλέπεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξέταση λοιπόν που κάνω σήμερα της κατάστασης όσον αφορά των εθνικών μειονοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά το 2015 και βασίζεται στον έλεγχο της εφαρμογής της σύμβασης πλαισίου. Και για να υπάρχει διαφάνεια πρέπει να σας πω ότι εγώ ίδια είμαι μέλος της ομάδας ελέγχου της εμβουλαστικής Επιτροπής της Σύμβασης αυτής εκ μέρους της Δανίας. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν θα αναφερθώ στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξετάστηκαν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή το 2014 και 2015 και όχι στις υπόλοιπες. Μιλάμε για 11 χώρες. Δεν είναι... Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί όλες οι απόψεις γιατί ακόμα βρισκόμαστε σε διαδικασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αλλά αν θέλετε μπορώ να σας δώσω περισσότερες ε, λεπτομέρειες. Επίσης, δεν θα μιλήσω τόσο για τους Ρωμά, γιατί υπάρχουν άλλοι συναδέλφοι που θα αναφερθούν σε αυτούς. Συνεπώς, η κατάσταση όσον αφορά τις εθνικές μειονότητες και την προστασία τους. Έχει να κάνει με δύο σκέλη. Το ένα είναι η έλλειψη της πολιτικής βούλησης και η αδράνεια των κυβερνήσεων όσον αφορά την προστασία των μειονοτήτων και δεύτερον έχει να κάνει με το πολιτικό κλίμα το σημερινό που έχει σαν αποτέλεσμα να ανέρχονται ακροδεξιά κινήματα με μια ατζέντα υπέρ της ξενοφοβίας και του μίσους. Όσον αφορά τον έλεγχο που κάναμε, διαπιστώσαμε ότι έχουμε διάφορες προδιαγραφές. Υπάρχει η ελευθερία όσον αφορά την αυτοαναγνώριση, ε, το δικαίωμα να αποφύγει κανείς την εφομία, να διατηρήσει τον πολιτισμό του, να έχει πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης, να μπορεί να χρησιμοποιεί γλώσσες μειονότητας και να τις χρησιμοποιεί στην επαφή του με τις δημόσιες αρχές, το δικαίωμα στη διγλωσία στο δημόσιο χώρο, το δικαίωμα να μαθαίνει γλώσσες μειονοτήτων και να έχει ευκαιρίες να διδαχθεί σε τέτοιες γλώσσες μειονοτήτων και το δικαίωμα συμμετοχής σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τη ζωή των μειονοτήτων. Αυτά είναι οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην σύμβαση πλαίσιο που οι περισσότερες χώρες έχουν ε, υπογράψει. Θα αναφερθώ σε μερικές περιπτώσεις μόνο. Τα υπόλοιπα υπάρχουν έτσι κι στην έκθεση που σας έχω υποβάλει. Παρά τις βελτιώσεις που έχουν ε, γίνει όσον αφορά την ισότητα και δεδομένου ότι υπάρχουν και μέτρα κατά των κρίσεων, παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της μένουν πολύ πίσω, δεν έχουν τους θεσμούς οι οποίοι χρειάζονται για να προστατεύσουν, να εφαρμόσουν δηλαδή αυτά τα μέτρα και να προστατεύσουν τις εθνικές μειονότητες. Ακόμα και αν υπάρχουν σώματα που ασχολούνται με την ισότητα, παρόλα αυτά δεν έχουν την ικανότητα, δεν έχουν αρκετό προσωπικό για να βοηθήσουν τους ε, αρμόδιους να αντιμετωπίσουν ζητήματα μειονοτήτων. Μια άλλη πτυχή είναι η ικανότητα αντιμετώπισης. Χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση, δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό για να αντιμετωπίσει όλες τις προσφυγές. Κάποια θέματα, ειδικά εξάλλου για τις μειονότητες, δύσκολα αξιολογούνται όπως το καθεστώς των θυμάτων πολέμου ή των ε, ανθρώπων που επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους. Υπάρχουν και πολλαπλές επίσης ε, διακρίσεις σε βάρος μειονετήτων, πολλές φορές και εξαιτίας φέλου και εξαιτίας ε, προσανατολισμού σεξουαλικού ή και αναπηρίας. Πολλές φορές υπάρχουν και τα τρία, γι' αυτό μιλάμε για πολλαπλές διακρίσεις. Πολύ λίγες ευρωπαϊκές χώρες δυστυχώς συλλέγουν στοιχεία για τέτοιου είδους διακρίσεις, οπότε χωρίς στοιχεία πώς θα τα καταφέρουμε. Το θέμα τώρα της προστασίας του πολιτισμού. Πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα στις γλωσσικές και εθνικές μειονότητες να διατηρούν και να αναπτύσσουν τον πολιτισμό τους. Εδώ έχουμε να κάνουμε κυρίως με τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτά αναφέρονται στην ε, σύμβαση πλαίσιο. Θα έπρεπε να υπάρχουν θετικά μέτρα, αλλά αυτά που ε, απαιτούν και οικονομική στήριξη. Αλλά μετά την οικονομική κρίση η τάση είναι το αντίθετο. Περικοπές στις δαπάνες για πολιτιστικούς οργανισμούς μειονοτήτων. Επίσης υπάρχει τάση να αποκλείονται μειονότητες από την λήψη αποφάσεων σε θέματα που έχουν να κάνουν με πολιτιστικές ε, πολιτικές. Και δεν υπάρχει και διαφάνεια, οπότε δύσκολα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οικονομικού πόρου οι μειονότητε. Οι κυβερνήσει θα πρέπει να είναι πιο ανοιχτέ και να περιλαμβάνουν και τι μειονότητε και τους τόπους που είναι σημαντικοί για τις μειονότητες να τους συμπεριλαμβάνουν στους επίσημους καταλόγους πολιτιστικής κληρονομιάς. Έρχομαι τώρα στις γλώσσες μειονοτήτων. Ένα σημαντικό θέμα για την προστασία της ταυτότητας των μειονοτήτων είναι το δικαίωμα της εκπαίδευσης στην γλώσσα των μειονοτήτων και με τον σχετικό πολιτισμό. Αυτό αναφέρεται ρητά στην σύμβαση πλαίσιο. Οι κυβερνήσει πρέπει να διασφαλίσουν επίσης τους κατάλληλου πόρου και ευκαιρίε ώστε να υπάρχει ισότητα στην εκπαίδευση. Πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευση και σε όλες τις γλώσσες των μειονοτήτων. Τέτοια προγράμματα αρχίζουν να γίνονται ο κανόνας στις περισσότερες χώρες μέλη αλλά εξαιτία της κρίσης δυστυχώς αυτό περιορίζεται τώρα. Έχουν, υπάρχει μείωση στη χρηματοδότηση, λιγότεροι δάσκαλοι στις γλώσσες μειονοτήτων, λιγότερο υλικό. Επίσης συγχωνεύονται σχολεία μειονοτήτων. Κάτι το οποίο έχει επηρεάσει κυρίως μειονότητες που ζουν σε απομακρυμένες περιοχές. Οι κυβερνήσεις δεν προστατεύουν τα μικρά αυτά σχολεία. Σε πολλές χώρες μάλιστα δεν έχουν στη διάθεσή του σύγχρονη τεχνολογία. Και όμως θα έπρεπε να μαθαίνουν τη δικιά τους γλώσσα μειονοτήτων. Όμως υπάρχει τάση να μαθαίνουν την γλώσσα της χώρας στην οποία ζουν και όχι τη δικιά τους μειονότητα, επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί καθηγητές. Δεν υπάρχει ένταξη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολλές φορές μιλάμε για ένα διπλό σύστημα που όμως μένει να ελεγχθεί. Οι, μειον... Οι μειονότητας λοιπόν Οι πολλές φορές οι άνθρωποι που έρχονται από μειονότητες γίνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας, κάτι που δεν βοηθάει στη συνοχή. Και έτσι έρχομαι στο δεύτερο σημείο που ανέφερα πριν, που έχει να κάνει με το σημερινό πολιτικό κλίμα, το οποίο επιτρέπει να υπάρχει μια τζέντα ξενοφοβίας και μίσους. Στην σύμβαση πλαίσιο αναφέρεται η ευθύνη των κυβερνήσεων σε δύο άρθρα. Στο 6 που μιλάει για την ευθύνη των κυβερνήσεων να προωθήσουν το διαπολιτισμικό διάλογο και για την αμοιβαία, τον αμοιβαίο σεβασμό, κάτι το οποίο δυστυχώς λείπει. Και υπάρχει και το άρθρο 12, όπου αναφέρεται στην υποχρέωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της ε, προστασίας του διακοινωτικού διαλόγου στις κοινωνίες. Σύμφωνα με τη σύμβαση πλαίσιο υπάρχει ευθύνη από τις κυβερνήσεις να ελέγξουν ότι όντως υπάρχει αυτός ο διαπολιτισμικός ε, διάλογος και την ευθύνη την έχουν οι κυβερνήσεις. Ο διάλογος αυτός πρέπει να υπερέχει παντού, σε όλες τις χώρες. Γιατί έτσι προστατεύονται τα δικαιώματα των ε, μειονοτήτων, αλλά προστατεύουμε και την ασφάλειά τους, γιατί δυστυχώς με τα ξενοφοβικά κινήματα πολλές μειονότητες, η Ρώμα για παράδειγμα, έχουν ε, περάσει από τη ρητορική μίσους, η οποία δυστυχώς δεν είναι αυξανόμενη. Η Ισλαμοφοβία, ο αντισημιτισμός επίσης πλήττουν τις μειονότητες και άλλες μειονότητες εκτός από τις καθ' Μία πτυχή προστασίας μειονοτήτων είναι η υποχρέωση μέτρων υπέρ της αμοιβαίας αναγνώρισης και κατανόησης για να προστατεύουμε από εχθρικές πράξεις και βιαιότητες τις μειονότητες αυτές. Όταν Επίση, συζητάμε για προσλήψεις στην αστυνομία. Πρέπει και οι μειονότητες να έχουν πρόσβαση. Δυστυχώ οι κυβερνήσει δεν το φροντίζουν αυτό. Οι πολιτικές εκπαίδευση επίσης δεν φροντίζουν για την διάδοση, την ενημέρωση για τις μειονότητες, τον πολιτισμό τους και τη γλώσσα τους. Ούτε καν τα μέσα ενημέρωση δεν το κάνουν αυτό. Τα βιβλία τη ιστορία δεν είναι αντικειμενικά πολλέ φορέ και δεν επικεντρώνονται στο διάλογο. Τα μέσα ενημέρωσης είναι μια μεγάλη ανησυχία για μας γιατί μπορεί κανείς εύκολα να έχει πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης. Το profiling επίσης από την αστυνομία είναι κάτι που ανησυχεί σε πολλές χώρες και ακόμα και αν υπάρχουν κανόνες οι κυβερνήσεις δεν εφαρμόζουν αυτούς τους, αυτούς κανόνες με συνέπεια. το χειρότερο είναι όταν δεν εφαρμόζουν καν την, ε, τέτοιους κανόνες στην νομοθεσία τους. Και για να καταλήξω, αυτή η σύντομη εξέταση των ανησυχιών μας όσον αφορά την προστασία των μειονοτήτων έγινε το 2014 και 2015 και δείχνει ότι δεν είναι ισότιμη η προσέγγιση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου δεν έχουν υπογράψει όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το καθεστώς για την προστασία των μειονοτήτων και όσες το έχουν υπογράψει μένει να κάνουν ακόμα πολλά για να το υλοποιήσουν. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει περισσότερα, παραμένει παρατηρείται επειδή δεν έχει τις αρμοδιότητες από την νομοθεσία που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, ε... Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Μαλόη. Ε, Ιβάνοφ τώρα. Ο κύριος Ιβάνοφ έχει, οργανω... έχει εργαστεί στην Βουλγαρία ως συνήγορος για πέντε χρόνια και έφερε πολλές υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενέπιου, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε εθνικά δικαστήρια σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και έχει περάσει και δύο χρόνια ως νομικός ε, σύμβουλος για θέματα ε, του προγράμματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σόφια της Βουλγαρίας. Τώρα εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα του Ρώμα. Ε, Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για τους Ρωμά, μια μειονότητα που δεν είναι και η μεγαλύτερη στην Ευρώπη το αέριο ως Ευρωπαϊκό Γραφείο Πληροφόρησης για τους Ρωμά είναι ευρέως ε, αναγνωρισμένο ε, γιατί έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση πολιτικών που εντάσσουν τους Ρωμά. Οι στρατηγικές ε, ξεκίνησαν πριν από 4,5 χρόνια με την έγκριση από την Κομισιόν αυτής της ε, επίσημης και γνωστής στρατηγικής. Τα ε, δικαιώματα των Ρωμά λοιπόν είναι και γραμμένα στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως είναι ευρέως δια γνωστό ότι υπάρχει, ε, υπάρχουν διακρίσεις, υπάρχουν διαχωρισμοί και γενικά ε, υπάρχει μεγάλος ε, αντιτσιγκανισμός ε, στον γενικότερο πληθυσμό. πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρωμά στις ανατολικές χώρες και τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Ε, όμως και οι Ρωμά που ζουν στη Δυτική Ευρώπη βιώνουν παρόμοιες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Παρά τις δεσμεύσεις ε, και τους πόρους που δίνονται, η κατάσταση στο Ρωμά λίγο έχει βελτιωθεί, αν έχει βελτιωθεί τα πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια. Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση των αντιτσιγκανικών συναισθημάτων σε κάποιες χώρες ε, που υποδαβλίζονται σχετικά ε, από τις διάφορες μορφές ε, που λαμβάνει η μετανάστευση κατά καιρού και ειδικά των Ρωμά. Το Ευρωπαρόμετρο του 2012 δείχνει ότι τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους συμφωνούν ότι ε, υπάρχουν αντιτσιγκανικά αισθήματα. Βέβαια, συνήθως ε, λέμε ότι οι έρευνες υπερβάλλουν, όμως το ευρωβαρόμετρο είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπα ότι βάσει αυτού τρεις στις τέσσερις Ευρωπαίους θεωρούν ότι οι Ρώμα αποτελούν αντικείμενο διακρίσεων και ότι ε, όλοι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πιστεύουν, το 34% των πολιτών θεωρούν ότι δεν είναι άνετοι όταν υπάρχουν Ρωμά παιδιά στα σχολεία των παιδιών τους ε, και όταν έχουν γείτονε που είναι Ρωμά ή εν μέρη Ρωμά. Πολλές ε, εκθέσεις επιστούν την προσοχή στην αποτυχία των πρωτοβουλίων που δεν είχαν συντονισμό, στην έλλειψη συμμετοχής των Ρωμά στη λήψη των αποφάσεων, στην ανεπάρκεια της νομοθεσίας, να αντιμετωπίσει τον αντιτσεκανισμό και άλλους ε, τέτοιους παράγοντες. Ε, που πρέπει να τους δούμε από νέα οπτική γωνία. Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και όταν υπάρχουν τα κονδύλια, υπάρχει συστηματική, υπάρχουν συστηματικές διακρίσεις που αποτελούν τη ρίζα των οικονομικών, κοινωνικών και άλλων πολιτισμικών προβλημάτων ανέχειας και αποκλεισμού των Ρωμά. Ε, συμφωνούν όλοι λοιπόν ότι για να υπάρξει βιώσιμη πρόοδος και βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρωμά πρέπει να ε, μειωθεί ο αντιτσικανισμός σε όλη την Ευρώπη δραματικά και σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες που συνεχώς, στις οποίες συνεχώς τα πάθη υποδαβλίζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους πολιτικούς κτλ. Τα στερεότυπα, τα ρατσιστικά, συνήθως ε, ενισχύονται ας πούμε με τις ε, επιχειρήσεις της αστυνομίας, τους καταπλησμούς των Ρωμά που είναι εντός εισαγωγικών εγκληματικοί κτλ. Επίσης, ε, ο αντιτζικανισμός ε, οδηγεί στην, ε, στο να εμποδίζει την εφαρμογή μέτρων που θα βελτιώσουν την κατάσταση των Ρωμά, ας πούμε, σε εθνικό επίπεδο έχουμε μόνο κοινέ υποσχέσεις που δεν εφαρμόζονται λόγω του πολιτικού κόστους. Θα έλεγα ότι ε, ένας από τους τρόπους που εκδηλώνεται η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρωμά είναι ο διαχωρισμός των Ρωμά από την υπόλοιπη κοινωνία. Η βελτίωση της στέγασης, της εκπαίδευσης, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη χωρίς να αντιμετωπιστεί το θέμα του διαχωρισμού, ε, μόνο βραχυπρόθεσμη λύση δίνει. Είναι σημαντικό λοιπόν να τονίσουμε ότι θελημένος αυτός διαχωρισμός στα σχολεία σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρόσφατα ξεκίνησε διαδικασία επιπαραβάση για την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία μια άλλη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κοινή έκθεση του 2014 για την εφαρμογή της ε, ε, οδηγίας ε, για τις, τη φυλετική ισότητα, αναφέρει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, όπως για παράδειγμα η έλλειψη ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα, έλλειψη στοιχείων για την ισότητα, μικρή ε, καταγραφή στοιχείων, ε, προβλήματα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, λίγες ε, κυρώσεις και ένδικα μέσα. Πολύ συχνά λοιπόν όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις πολλαπλών διακρίσεων συνήθως οι νομοθέτες δεν έχουν στοιχεία για να βρουν τις λύσεις. Το πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με την Κομισιόν, σπάνια προέρχεται άμεσα από την νομοθεσία, αλλά από την εφαρμογή της. Έτσι λοιπόν ε, θέλουν στην Κομισιόν να περάσουν τον έλεγχο ε, και στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Αυτό ακριβώς αναφέρεται σε αυτή την τελευταία έκθεση. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει και να εφαρμόσει πιο στεναρά τις πολιτικές και την ομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα, γιατί ε, η Ρωμά είναι από τις πλέον ε, μειονεκτικού πληθυσμού στην Ευρώπη και θα είναι οι πρώτοι που θα υποφεληθούν από αυτέ τι πολιτικέ Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη το ε, αντίκτυπο των διαφόρων γεωπολιτικών εξελίξεων στην εφαρμογή των ατζέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα. Η αύξηση τη ακροδεξιά, των εθνικιστικών τάσεων στην Ευρώπη, η αύξηση των μέτρων για την ασφάλεια και κατά τη τρομοκρατία αποτελούν άμεση, ε, έχουν, και οι κρίση των προσφύγων έχουν άμεση σχέση με την παραβίαση των βασικών δικαιωμάτων γενικότερα ε, και με την εφαρμογή ε, των πολιτικών για την ενσωμάτωση των Ρωμά και την ίση μεταχείρισή τους. Έτσι λοιπόν η ε, μάχη κατά του κρατεού αντιτσιγκανισμού απαιτεί αιμονή και αποφασιστικότητα. Το πρώτο στάδιο είναι να αναγνωρίσουν οι δημόσιοι λειτουργοί ότι υπάρχει αυτή η τάση και να ε, καταδικάσουν κάθε εκδήλωσή της επιπλέον. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ένα ρόλο να παίξουν Πρέπει να υπάρξουν εκστρατείε ε, να υπάρχει εκπαίδευση κατά του ρατσισμού, ε, ειδικά των ερετών, των δημοσίων υπαλλήλων της αστυνομίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των ε, δασκάλων και των κοινωνικών λειτουργών. Η οργάνωσή μου είναι το μεγαλύτερο δίκτυο Ρωμά στην Ευρώπη και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τι Εθνικέ αρχέ και την κοινωνία των πολιτών, επικεντρώνοντα το ενδιαφέρον σε βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ε, πολιτική σε τομεακό επίπεδο που θα προωθήσει ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την συμμεταχείριση των Ρωμά και άλλων μειονεκτικών ομάδων. Υπάρχουν ε, τα μέτρα που μπορούν να πατάξουν τι συνεχεί διακρίσει, τα μέτρα που θα αντισταθμίσουν τι προηγούμενε διακρίσει διακρίσεις και αυτά που θα μειώσουν τις ε, ε, διακρίσεις στο μέλλον. Σύμφωνα με ένα άλλο ε, στοιχείο του Ευρωμαρόμετρου υπάρχει μια άλλη μορφή διακρίσεων, αυτή που βασίζεται στην εθνότητα, τα 64%. Η βία όμως που προέρχεται από αυτές τις διακρίσεις δεν αντιμετωπίζεται από τις αρχές. Οι ε, διακρίσεις ε, γίνονται όλο και πιο θεσμο, θεσμοθετούνται όλο και περισσότερο. Υπάρχει ρητορική μίσους που καθημερινά ακούγεται και εκφράζεται ξεκάθαρα και ελεύθερα στα εθνικά κοινοβούλια από τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων, των, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ε, είναι κάτι που βλέπουμε συνεχώς γύρω μας και μας γύρει κάποια ερωτήματα σχετικά με το πώς θα προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ε, ισότητα ως βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση απαιτεί επίγουσα δράση από τους θεσμούς και την κοινωνία των πολιτών. Όπως είπε και ο καθηγητής πριν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ιβάνοφ, ο κύριος Ιβάνοφ, μάλλον πρέπει να φύγει σύντομα, οπότε αν υπάρχει κάποια ερώτηση για αυτόν τώρα, για τον κύριο Ιβάνοφ. Δεν υπάρχει ερώτηση. Ωραία, καλώς. Εντάξει κύριε Ιβάνοφ, σας ελευθερώνουμε συνεπώς. Πολύ ενδιαφέρον όσο μας είπατε. Ο επόμενος είναι ο κύριος Κάτας, ο οποίος έχει ιδρύσει από κοινού με άλλους την οργάνωση, τη Διεθνή Οργάνωση για τα άτομα ακαθόριστου φύλου. Το 2013 έγραψε ένα βιβλίο που αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ των φύλων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την Επιτροπή σας που μας κάλεσε για να έρθουμε να σας μιλήσουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα καθόριστου φύλου, μεσοφυλικοί όπως ονομάζονται. Ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα για να αρχίσουμε διάλογο με το μεταξύ τα άτομα αυτά γεννιούνται με κύριε και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά φύλου, όπω είναι τα εσωτερικά και τα εξωτερικά γενετικά του όργανα, χρωμοσώμα, γενετήσια δένε, ορμόνε, μυϊκή μάζα, κατανομή τριχωτού, σωματική διάσταση, που είναι χαρακτηριστικά που δεν ανήκουν μόνο στου άντρε ή στι γυναίκε ή μπορεί να ανήκουν και στα δύο. Κάποιε παραλλαγή χαρακτηριστικών φύλου όμω από τον ανδρικό κόσμο θεωρούνται ω δυσλειτουργή για την ανάπτυξη του φύλου. Μια τέτοια διάγνωση συχνά συνοδεύεται και από την έννοια ότι το άτομο αυτό πρέπει να διορθωθεί με ιατρική βοήθεια. Για το να διορθώσουμε εντό αγωγικών ένα τέτοιο άτομο σημαίνει ότι θα το υποβάλουμε σε θεραπεία για να αλλοιώσουμε τα χαρακτηριστικά του φύλου του μέσω χειρουργικών επεμβάσεων ή ορμονικής ε, θεραπείας. Αυτό σημαίνει επίση ότι έτσι οι άνθρωποι αυτοί θα ανταποκρίνονται καλύτερα στι προσδοκίε τη κοινωνία, όσον αφορά δηλαδή τα χαρακτηριστικά του πραγματικού του φίλου έτσι όπως το θέτει η ιατρική κοινότητα. Το 2014 έγινε μελέτη από το Ολλανδικό Ινστιτούτο για Κοινολογικές Έρευνες που σύγκρινε τα στοιχεία και βρήκε ότι ένα στα 200 άτομα είναι μεσοφιλικό. Δηλαδή ένα στα 200 άτομα σύμφωνα με τον ιατρικό κόσμο χρειάζεται ιατρική φροντίδα για να διορθωθεί. Υπάρχουν ηθικές επιπτώσεις όπως καταλαβαίνετε και όχι μόνο. Ε, γίνονται πολλές φορές ε, διαγνώσεις για τέτοιες περιπτώσεις ακόμα και σε επίπεδο προεμφύτευσης. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα είναι ότι για να αποφύγουμε την παραλλαγή τέτοιων ε, χαρακτηριστικών οδηγούμαστε σε άμβλωση, σε προχωρημένο στάδιο πολλές φορές. Το αποτέλεσμα όμως από τις διάφορες παρεμβάσεις έχουν σαν αποτέλεσμα να ακολουθούνται διάφορες ε, πρακτικές από ακροτηριασμό στην κλειτορίδα, φέρεση, από κολποπλασία, ε, κολπική διαστολή, αλλάζει το σημείο που βρίσκεται η ορίθρα, τοποθετείται ε, αλλού κτλ. Σύμφωνα με το 2015 πάντως και τον ΦΡΑ, παραβιάζονται έτσι τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αυτών. Όμως παρόλα αυτά ε, ακόμα προτείνονται χειρουργικές επεμβάσεις και πολλές φορές σε πολύ νωρί ηλικία, δηλαδή τα πρώτα δύο χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Σε οχτώ χώρες μέλους ένας νομικός εκπρόσωπος πρέπει να συνενέσει ανεξάρτητα από την ικανότητα του παιδιού να αποφασίσει από πόνο του ή όχι. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει αυτοδιάθεση αλλά υπάρχει παραβίαση αυτή τη αρχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σεβόμαστε τη φυσική και ψυχική ακαιρεότητα όλων. Ιατρικές θεραπείες, χωρίς να έχει συμφωνήσει απόλυτα το διαφερόμενο άτομο, είναι παραβίαση του δικαιώματος στην φυσική και ψυχολογική ακαιρεότητα, ενώ αναφέρονται οι αρχές αυτές στα δικαιώματα των ατόμων στο άρθρο 3 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και στα δικαιώματα για το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, στο άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κλπ. Οι παρεμβάσεις αυτές επίσης αποτελούν απάνθρωπη θεραπεία και υποβιβαστική σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη και τον ειδικό εισηγητή για τις ε, για τα βασανιστήρια. Όταν ε, γίνονται τέτοιες ε, παρεμβάσεις γίνονται συνήθως από την παιδική ηλικία. Τι γίνεται με τους ενήλικες, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν περάσει από τέτοιες ιατρικές και ψυχολογικές παρεμβάσεις τις τελευταίες ε, πέντε δεκαετίες. Στιγματίζονται, βρίσκονται υποδιάκριση, παρενοχλούνται, δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική θεραπεία ή πρόσβαση σε ιατρική θεραπεία όπως χρειάζεται, δεν αναγνωρίζονται νομικά και κάπου είναι και όρατοι. Δεν υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση επίσης. Αναγκάζονται να φύγουν συχνά από το σχολείο. Δυσκολεύονται με ένα σωρό τρόπους, χάνουν την αυτοεκτίμησή τους. Τα άτομα αυτά δεν εκπροσωπούνται και πουθενά. Οι παραλλαγές των χαρακτηριστικών αυτών των φύλων δεν συμπεριλαμβάνονται σε κανένα σχολικό πρόγραμμα. Όταν μεγαλώνουν τα άτομα αυτά και γίνονται ηλικιωμένοι χρειάζονται πολύ περισσότερο πρόσβαση στην υγεία. Όμως η πρόσβαση στη γενική υγεία συχνά είναι πολύ πιο δύσκολο για τα άτομα αυτά εξαιτία ασφαλιστικών πρακτικών. Έτσι παραβιάζεται το δικαίωμά τους βάσει του άρθρου 35 της Ευρωπαϊκής Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, όπως το να κάνουν προληπτικά check-ups, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν συχνά με τη δήλωση του φίλου. Άλλα θέματα που αντιμετωπίζουν τα μισοφιλικά άτομα είναι ότι δεν έχουν πρόσβαση σε ορμονική υποκατάσταση, τουλάχιστον αυτοί που πραγματικά χρειάζονται τα άτομα αυτά, αντί να αλλάξουν φύλο. Από το 2008 οι χώρες μέλη έχουν ζητήσει πολλές φορές, έχουν, ο ΙΕ έχει ζητήσει από πολλές χώρες μέλη να πάρουν νομοθετικά και άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν το σεβασμό της φυσικής ακαιρεότητας και της αυτονομίας των ατόμων ακαθόριστου φύλου και να διασφαλίσουν ότι κανεί δεν θα περάσει από άχρηστε ή μη αναγκαίες οι ιατρικές διαδικασίες, ούτε όταν είναι παιδί, ούτε αργότερα. Το 2015 ο Επίτροπος για Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου τη Ευρώπη δημοσίευσε ένα έγγραφο για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων αυτών. Τα σώματα των Ηνωμένων Αθνών, όπως επίσης και το CHRCOE, πιέζει τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ε, οι υπηρεσίες συμβουλών προς τα άτομα καθόριστου φίλου και τους γονείς τους. Να φροντίσουν πάντα ότι πρέπει να δίνουν τη συνένεσή τους τα άτομα αυτά προκειμένου να περάσουν υποτρική θεραπεία ή χειρουργείο. Να ε, περιμένουν τη στιγμή που πρόκειται για μη αντιστρεπτές ε, πρακτικές να μεγαλώσουν τα παιδιά για να μπορούν τα ίδια να δώσουν τη συνένεσή τους. Επίσης, να υπάρχει βοήθεια για την φυσική και ψυχολογική πίεση που υφίστανται τα άτομα αυτά. Μέχρι τώρα, μόνο η Μάλτα από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν απαγορεύσει τη μη συνενητική ιατρική παρέμβαση και ακολούθησε και η Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2015 με ένα νόμο κατά των διακρίσεων εξαιτία χαρακτηριστικών φύλου. Δυστυχώς όμως, γιατί εμείς θέλουμε να πιέσουμε την Επιτροπή σας να πιέσει, να υποφελθεί από αυτή την ευκαιρία για να υπάρξει μεγαλύτερη συνδυτοποίηση για τα άτομα καθόριστου του φύλου. Οι προτεραιότητες μας είναι να απαγορεύεται η ιατρική θεραπεία επί των ατόμων αυτών χωρίς τη συνένεσή τους, χωρίς να μπορούν ελεύθερα να αποφασίσουν γι' αυτό. Η νομοθεσία κατά των διακρίσεων επίσης να περιλαμβάνει και τα άτομα με παραλλαγές χαρακτηριστικών φύλου, προκειμένου τα άτομα αυτά να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να αποφελούνται των δικαιωμάτων τους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια συγκριτική μελέτη επίσης χρειάζεται όσον αφορά τις πρακτικές αυτές και να περιλαμβάνονται οι παραλλαγές του φύλου. Μια έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρει τη θέση του Κοινοβουλίου για τα άτομα αυτά είναι ευπρόσδεκτη. Θα πρέπει να πάρετε στα χέρια σας την ευθύνη για να βοηθήσετε τα άτομα αυτά να ζήσουν καλύτερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Thank you, uh, uh, Mr. Gattas. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκάτας. Επόμενος ε, ε, ε, ο μιλητής, ο κύριος Πατ Κλάρκ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Φόρουμα για την Αναπηρία και ε, αυτή τη στιγμή λαμβάνει μέρος σε ανεξάρτητες ε, ε, πρωτοβουλίες για άτομα με σύνδρομο Down στην Ιρλανδία. Έχει λάβει μέρος σε κινητοποιήσεις που διασφαλίζουν ότι τα άτομα με σύνδρομο Down και νοητική στέρηση έχουν μία πρόσβαση στις, σε όλες τις υπηρεσίες. Κύριε Κλάρκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με χαρά μου βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μιλήσω σε αυτή την πολύ σημαντική συνεδρία εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αναπηρίας που είναι ένας οργανισμός ομπρέλα που εκπροσωπεί εθνικά συμβούλια άτομα με αναπηρία σε όλη την Ευρώπη, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και μια σειρά από ευρωπαϊκά ε, και εθνικέ οργανώσεις ε, που σχετίζονται μαζί μας και δεν είναι σήμερα εδώ. Είμαστε μια ενωμένη φωνή των ανθρώπων με αναπηρία στην Ευρώπη. Χαιρόμαστε που έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί σας για τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων σε αυτή εδώ τη δημόσια ακρόαση πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση από την πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία αναφέρονται στην Σύμβαση των Εθνών για τα άτομα με αναπηρία που δεν έχει που έχει κυρωθεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη. Δυστυχώς, η ε, χώρα μου η Ιρλανδία πόρα απέχει από μια καλή κατάσταση ε, σε αυτό το επίπεδο. Ε, ελπίζουμε να διορθωθεί αυτό μέχρι το τέλος του έτους. Είναι για άλλη μια φορά στην ιστορία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμευμένη λοιπόν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα προγράμματα, οι πολιτικές και οι αποφάσεις πρέπει να συνάδουν με αυτή τη σύμβαση. Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να ενσωματώνονται ως διάσταση σε όλες τις στρατηγικές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλες τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η νέα προσέγγιση λοιπόν απαιτείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διαμόρφωση των πολιτικών. Τελευταία ε, ήταν ε, πρόσφατα που έγινε ε, μία σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση το Σεπτέμβριο του 2015 συγκεκριμένα από τον ΟΗΕ ε, που δίνει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς θα προωθήσει, θα προστατεύσει και θα διασφαλίσει καλύτερα τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία στην Ένωση. Έχει μια λεπτομερή λίστα δράσεων και μέτρων που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Οι συστάσει δίνουν μια σειρά προτεραιοτήτων, ξεκάθαρη ένα οδικό χάρτη για τι δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, έτσι ώστε να εφαρμοστεί σωστά η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία και να προστατευτούν αυτά εντό της Ένωση. Οι συστάσει αυτέ ε, είναι το βασικό σημείο αναφορά για το μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον επόμενο μήνα θα υιοθετήσει ένα ψήφισμα με βάση αυτά τα συμπεράσματα. Και τις παρατηρήσεις ε, και είναι η ευκαιρία σας να αντιδράσετε. Θέλουμε να ευκράσουμε λοιπόν την ευγνωμοσύνη μας ε, στο Κοινοβούλιο και την κυρία Στίβενς ως εισηγήτρια γιατί έχει περιβα... λάβει τα άτομα με αναπηρία σε αυτό το ψήφισμα στις καταληκτικέ παρατηρήσεις, η Επιτροπή του Ηνωμένων Εθνών ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει διαρθρωτικό διάλογο με τα άτομα αυτά που εκπροσωπούνται από διάφορες οργανώσεις. Πρέπει όλες οι πολιτικές και λήψεις αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σχετίζονται με τη σύμβαση και να πάμε πέρα από τι ad hoc ε, καταστάσεις συμμετοχή ε, των ανθρώπων με αναπηρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντοτε ε, ο ηγέτης, ε, η πρώτη που κύρωσε. Τώρα πρέπει να είναι ε, αυτή που θα εφαρμόσει αυτό το πλαίσιο και πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική που θα είναι αφοσιωμένη σε αυτήν την σύμβαση. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αναπτυρία 2010-2020 Εγκρίθηκε πριν από τη σύμβαση και φέτος έχουμε απλώς μια αναθεώρηση. Δεν έχουμε ένα πραγματικό σχέδιο δράσης σε βάση της εφαρμογής αυτής της σύμβασης και αυτό με ανησυχεί. Υπάρχει μια ανησυχητική τάση να μην λαμβάνεται σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Από τη Γενική Διεύθυνση Justice πήγαμε στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για αυτό το θέμα. Η οδηγία για την ίση μεταχείριση, η οριζόντια οδηγία, <clears throat> έχει φέρει 60 εκατομμύρια ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και διακρίσεις λόγω θρησκευτικού, προσεξουαλικού προσανατολισμού, φιλετικής προέλευσης να γνωρίζουν διακρίσεις σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Χρειάζεται γρήγορη έγκριση τη πρόταση βάσει και των όσων προβλέπει η Σύμβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανταποκριθεί στην κρίση των προσφύγων δεν βασίστηκε σε μια προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ΔΕΕΦ ανησυχεί ιδιαίτερω για την κατάσταση των ανθρώπων με αναπηρία που μπορεί να φτάνουν στην Ευρώπη. Πρέπει να αναλυφθούν μέτρα για να γίνει η απόκριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην κρίση των προσφύγων και των μεταναστών και ε, συνολική και ε, συμμετοχική. Θα πρέπει να εφαρμοστούν οι καταληκτήριες ε, παρατηρήσεις μας η Επιτροπή συνέστησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει το ποσοστό απασχόληση στις πολιτικές της. Η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει τις κατευθυντήρε γραμμές που εξέδωσε και να μην επιτρέπει την κράτηση των ανθρώπων ε, με ειδικέ ανάγκες στο πλαίσιο τη μετανάστευση και τη αίτηση ασύλου. Όλα αυτά δεν συνάδουν με τη σύμβαση. Επιπλέον, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων με ειδικέ ανάγκε δεν έχουν νομικέ δυνατότητε, δεν έχουν δικαίωμα να προσφύγουν σε εθνικό επίπεδο. Οι αποφάσεις ε, για μερική ή συνολική κυδαιμονία των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκε μπορεί να μην γίνουν αποδεκτά. Ή και τα δικαιώματα που προβλέπουν οι συνθήκε και οι νομοθεσίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να, μην προβλέπουν, να μην προβλέπουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη, τι βασικέ υπηρεσίε όπω η τράπεζα, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη. Όπω και τα καταναλωτικά δικαιώματα ή τα, δικαιώματα του, ε, των δοσοληψιών. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα ξαναδεί αυτά με τα κρατημέλη. Επίση, η Επιτροπή ε, ζητά και την δημιουργία ενός ε, προτύπου για την ελάχιστη κοινωνική προστασία. Πρέπει η σύσταση αυτή να ακολουθηθεί, διότι τα άτομα με ειδικέ ανάγκε έχουν πληγεί ιδιαίτερω από τον περιορισμό των υπηρεσιών, ιδίω αυτών που του επιτρέπουν να ζουν ομαλά σε μια κοινότητα. Η υποβάθμιση ε, τη ποιότητα ζωή του ε, οφείλεται στην απομονωμένη δράση των θεσμικών οργάνων. Η Επιτροπή μα πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει και το ποσοστό απασχόληση στην αγορά εργασία και να αποτρέψει τα περισσότερα τι περαιτέρω συνέπειε των μέτρων λιτότητα. Πρέπει όλα τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων τα διαδοτικά και τα κονδύλια τη ΕΕ, να χρησιμοποιηθούν για να προωθήσουν την υλοποίηση τη σύμβαση στα κράτη-μέλη και στι τρίτε χώρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει με τα, ποσά, με τα να φροντίσει να μην οικοδομούνται απομονωμένα σχολικά ιδρύματα ή στεγαστικές ε, εγκαταστάσεις. Όλες οι πληρωμές που έχουν δοθεί κατά παράβαση τη σύμβαση αυτή πρέπει να ανακληθούν. Ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ε, το επιβεβαιώνει αυτό με μια πρόσφατη αποφασή του που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να χρηματοδοθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια δράσει που δεν συνάδουν με τι αξίε τη Ένωση. Δηλαδή τα δικαιώματα και τι ηλοφερίε καθώ και τι αρχέ που αναγνωρίζει η Χάρτα. <clears throat> Τέλο, η EDF καλωσορίζει την ε, δημοσίευση της ευρωπαϊκής ε, πράξης, νομικής πράξης για την προσβασιμότητα ως μια δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βελτιώσει την ε, πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους. Έχει τεράστιο δυναμικό αυτό για όλη την Ένωση και προστιθέμενη αξία για τα άτομα με αναπηρίες. Ε, ωστόσο, αυτή η πράξη Ε, εφόσον ανατεθεί στην ε, CRPD ως προς την εφαρμογή της, θα πρέπει να συνάδει με όλα τα κριτήρια της CRPD. Η πρόταση αυτή έχει κάποιες ε, λήψεις και κενά ως προς τον σεβασμό του άρθρου 9 της σύμβασης. Η διεύρυνση του πεδίου θα ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να βελτιωθούν, ώστε η πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες να γίνει πραγματικότητα. Για να ολοκληρώσω, Ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει ηγετική δράση στην υλοποίηση των ε, συστάσεών μας. Οι συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο φιλόδοξη και ε, προσεκτική στην υλοποίηση των συστάσεων της Σύμβασης. Ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να ακολουθήσει την ίδια φιλόδοξη και αφοσιωμένη προσέγγιση και θα συνεργαστούμε και με την ΕΔΕΦ e για να πετύχουμε την κοινά μας τα κοινώς επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Κλάρκ. Τελευταίος ομιλητής μας, η κυρία Νατάσα Καζατσκίν, συντονίστρια συντονίστρια για την ομάδα εργασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικτύου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατία και ανώτερη πολιτική αναλύτρια θεμελιωδών δικαιωμάτων, δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων στο Ίδρυμα τη Ευρώπη για την Ανοιχτή Κοινωνία και την Πολιτική τη. Έχετε το λόγο, κυρία Καζάτσικη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την ε, πρόσκληση να απευθυνθώ στην Επιτροπή σα, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών σήμερα. Όπω αναφέρθηκε, σήμερα παίρνω το λόγο εκ μέρου της μη κυβερνητική οργάνωσης HIDN που βασίζεται, έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες είναι μια ομάδα 20 με κυβερνητικών οργανώσεων που δρούν στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων το δίκτυο των σχετικών ανθρωπίνων ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων με την ανάλογη πλατφόρμα, με εμπειρογνωμοσύνη για το θέμα αυτό. Έχουμε ε, συγκεντρωθεί πριν από ένα χρόνο και έχουμε αρχίσει την κοινή μας δράση για να διευκολύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα προσθέσω περισσότερα όσα είπαν πριν συνάδελφοι στα δικαιώματα των μονοτήτων, όμως θα ήθελα να ολοκληρώσω το σημερινό πάνελ μιλώντας για τα ευρύτερα ευρωπαϊκά θεσμικά ε, ζητήματα μετά τις προηγούμενες παρουσιάσεις. Υπάρχουν κάποιε συστάσεις που αφορούν την κοινωνία των πολιτών, καθώς και η ανάγκη για μια εσωτερική ε, ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανθρώπινα δικαιώματα. Πριν από δύο μέρες, και αυτό το ανέφερε η Επιτροπή, η Επιτροπή οργάνωσε μια συνάντηση για την εκκίνηση του νέου, ε, της νέας ομάδας υψηλού επίπεδου για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και άλλων μορφών έλλειψη ανοχή μη κυβερνητικέ οργανώσει συμμετείχαν από την αρχή στην οργάνωση τη εκδήλωση και εκπροσωπήθηκαν την ίδια την στην ίδια την ημερίδα με ε, μεικτά και, ε, πάνελ και πάνελ επίδραση. Θα ήθελα να πω εδώ στην Επιτροπή σα ότι υπάρχουν θέματα πρωτοκόλλου και πρακτικά θέματα, αλλά όσο δυνατόν περισσότερο καλό θα ήταν να αποφεύγουμε να ε, συμμετέχουν μόνο με κυβερνητικέ οργανώσει ε, σε πάνελ όπω το σημερινό. Και κλείνω εδώ την ε, παρένθεση. Ε, υπάρχει μεγάλη ανησυχία μεταξύ των με κυβερνητικών οργανώσεων για τον συρρυκνούμενο χώρο που αφήνεται στην κοινωνία των πολιτών παντού αλλά ιδίω στην Ευρώπη. Έχουμε δει επανειλημμένε επιθέσει κατά των με κυβερνητικών οργανώσεων σε εκστρατείε του στην, Ουγγρανία, στην Ουγγαρία, την ε, Πολωνία και τη Λιθουανία. Περιορισμό τη ελευθερία του διαδηλώνει και τη ελεύθερη έκθεση στην Ισπανία, καθώ και κατάρρευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ω προ την προσφορά βοήθεια στου μετανάστε και πρόσφυγε που φτάνουν στα ελληνικά νησιά, λόγω χάρη. Επίση, μα ανησυχεί η υποβάθμιση τη δημοκρατική λογοδοσία με τι ταχείε κοινοβουλευτικέ διαδικασίε και η έλλειψη διαφάνεια αυτών. Λόγω χάρη, η προτινόμενη Ευρωπαϊκή Οδηγία για την καταπολέμηση τη θερμοκρατία που συζητείται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβουλίο σα υποβλήθηκε χωρί καμία μελέτη αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πέρασε πολύ γρήγορα και από το Συμβούλιο. Η φάση σύνταξη τη νέα πρόταση για το άσυλο ε, έγιναν όλε σε μυστικέ συνομιλίε και πολύ λίγα πράγματα δημοσιεύτηκαν στο τέλο. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει στήριξη και να έχει ε, μεστό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών ω ένα καθοριστικό στοιχείο των διαδικασιών λήψη αποφάσεων και χάραξη πολιτικών. Αυτό με ε, πλήρε διαβουλεύσει ώστε να έχουν το χρόνο και οι πρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών για να συνεισφέρουν, να υπάρχει κοινή κατάρτιση τη ατζέντα των συναντήσεων, καθώ και παρακολούθηση το πώ δρά η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε αν υπάρχουν αποτελέσματα και να ενημερώνεται για κοινή γνώμη. Αυτό δεν τονίστηκε αρκετά στι παρεμβάσει του πρώτου πάνελ, οπότε ήθελα πραγματικά να το υπογραμμίσω. Όπω είπε και ο ΙΕ, το να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον κατάλληλο για τι μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι πυλώνα οποιοδήποτε συστήματο που θα χτιστεί γύρω από το σεβασμό του κράτου δικαίου. Γι' αυτό η ομάδα μα ε, ζήτησε να υπάρξει τροποποίηση στη σχετική έκθεση και να αναγνωριστεί επισήμω ο ρόλο τη κοινωνία των πολιτών και του κράτου δικαίου σε οποιοδήποτε μηχανισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και σεβασμού του, καθώ και κριτήρια για την αξιολόγηση του σεβασμού του κράτου δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Επίση, καλέσαμε την ε, οργάνωση διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και αυτό να συμπεριλαμβάνεται και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου στην ε, για το θέμα τη χάρτας και της εξωτερική και εσωτερικής συνοχής τη πολιτική μας. Παρά την ανοιχτή και συμμετοχική υποτίθεται στάση της Ολλανδικής Προεδρία απέναντί μας, ήταν πολύτιμο αυτό, αλλά απογοητευτήκαμε εν τέλει. Διότι όλα αυτά τα λόγια τελικά δεν συμπεριληφθήσαν σε συμπεράσματα του Συμβουλίου. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή, ήθελα να καταγραφεί σήμερα στα πρακτικά ότι ω ομάδα έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαν για να συζητήσουμε μαζί του απευθεία τη συνολική του θεώρηση για τη στρατηγική του για την ενίσχυση της ε, δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω πρωταγωνιστού στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Και φτάνω στο δεύτερο σημείο για τη στατική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επικριτικό σχόλιο που ακούγεται πολύ συχνά και θέλω να επιμείνω σε αυτό. Η στρατηγική αυτή, όπως προτείνεται, δεν είναι κίνητρο για τη δημιουργία ε, ενό χάρτινου τίγρη ε, όπως ε, θα το έθετε ένας ε, Ευρωπαίος υπάλληλος ή ένας υπάλληλος του ΟΗΕ. Θέλουμε αποτελέσματα. Εμείς αυτό θέλουμε ως μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δράση. Όχι αφηρημένες και θεωρητικές συζητήσεις. Όχι, φτάνει. Θέλουμε πραγματιστική, ρεαλιστική προσέγγιση, γιατί έχουμε μακρά πείρα ω ε, υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέλουμε πραγματικά να υπάρξει ευρωπαϊκή δράση για το σεβασμό, την προστασία και κυρίω, αυτό το έθεσε ο κ. Δεσκούτερ, ε, κυρίω για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη σε συναντήσει υψηλού επίπεδου, αυτέ που ανέφερα προηγουμένω δηλαδή, αυτέ προδιημέρου, ένα συμμετέχον νομίζω σημείωσε και είναι ενδιαφέρον ότι εάν σκεφτεί κανεί όλη την εμπρογνωμοσύνη που διαθέτουμε στην αίθουσα από τα κράτη-μέλη, από τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, από τον ΟΗΕ, τον ΟΑΣΕ, το Συμβούλιο τη Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε διεξοδικότατο, σφαιρικότατο σύστημα ε, και μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη βία που έχει υποδαπλιστεί από εκφράσεις η πρόκληση είναι πώς θα ε, κάνουμε αυτές τις εμπειρίες να ε, ε, γίνουν γνωστές σε όλους ταυτόχρονα. Να υπάρξει διαλειτουργικότητα. Υπάρχουν πόροι, αλλά πρέπει να διατεθούν ταυτόχρονα. Η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να γίνει πρωταρχικό στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει αυτό κάπου να δηλωθεί επισήμω και όταν συντονίζει τις προσπάθειες των κρατών μέσα των τριών θεσμικών οργάνων και σε όλε τι πολιτικέ τη. <clears throat> σε ό,τι αφορά τον συντονισμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο πώ η Επιτροπή και το Συμβούλιο στι πρωτοβουλίε του για την προώθηση του κατώτατου δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν συμβαδίσει πουθενά. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χαράξει μια εσωτερική διαδικασία για την παρακολούθηση και την ε, επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον σεβασμό του στο στο εσωτερικό των κρατομελών με το πολωνικό προηγούμενο, ε, το Συμβούλιο έχει σχεδιάσει κάτι τελείω διαφορετικό με μια πλήρω πολιτική συζήτηση. Η τελευταία πρόταση ε, της Ολλανδικής ε, Προεδρία έχει να κάνει με την ανταλλαγή μυστικών πληροφοριών στην Ευρώπη. Δεν έχει συνδυαστεί αυτό όμω με την εξελισσόμενη δουλειά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε με όλε τι ευρωπαϊκέ νομοθετικέ πράξει που συζητιούνται ούτε με τι προτάσει για το σύστημα ασύλου. Αυτό στέλνει ε, μηνύματα λίγο ε, περίεργα, μπερδεμένα για τις προτεραιότητε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το πώς ε, μπορεί να έχουμε έναν να έχουμε καλά αποτελέσματα από αυτέ τι μεμονωμένε προσπάθειε. Θέλουμε λοιπόν και στο σχέδιο έκθεση Ιντβελ αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο να παραλάβει την έκκληση για ενισχυμένο, εντατικότερο διάλογο μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων τη Ένωση. Ελπίζουμε αυτό να τονιστεί και πάλι στην ε, επικείμενη έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίση, να καλωσορίσουμε εδώ την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου να κατονομάσει ο κράτη όταν αυτό είναι απολύτω αναγκαίο, για να ε, είναι στοιχειοθετημένη η δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφέρομαι στην στο ψήφισμα τη CIA τη περασμένη εβδομάδα και το ψήφισμα για την Ουγγαρία. Αυτό θα πρέπει να γίνεται συστηματικότερα. Οπουδήποτε δει και δεν είναι πάντοτε έτσι στι εκθέσει για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και σημειώνω εδώ ότι στην έκθεση τη Επιτροπή για την Χάρτα δεν υπάρχει καμία ε, συγκεκριμένη γραμμή γι' αυτό. Κάποια κάτι αναφέρονται, αλλά τυχαία. Ω προ την παρέκκληση του από το κεκτημένο του ασύλου, κάποια άλλη όχι. Όταν μιλάμε για τη διακριτική μεταχείριση κατά τον Ρωμά. Για να πετύχουμε καλύτερη θεσμική συνεργασία και σκοπιμότερη δράση των θεσμικών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει όλες οι αποφάσεις να θεμελιώνονται κάπου. Αυτό είναι η ουσία τη στρατηγική μα. Πρέπει να υπάρχει κατανομή τη ευθύνη, τη συλλογική ευθύνη. Αν θέλουμε να πετύχουμε αλλαγή στην πράξη και εφόσον βασιζόμαστε σε κοινού ανθρωπιστικού στόχου, οι οποίοι ορίζονται από το διεθνέ, ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο. Είναι ο μόνο τρόπο να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει συνεκτική και αποτελεσματική δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να υπάρξει και προστιθέμενη αξία στι διεθνεί, εθνικέ και τοπικέ προσπάθειε. Να δώσω κάποια παραδείγματα του πως δεν υπάρχει ακόμη αρκετή διασύνδεση μεταξύ των προσπαθειών στην πράξη. Και θα αναφερθώ και πάλι στη συνάντηση προδιημέρου για την ρατσιστική βία και άλλες μορφές διακριτικής μεταχείρισης. Οι φρικαλες επιθέσεις στο Ορλάντο καταδικάστηκαν ομόφωνα στη συνάντηση. Όμως ούτε η Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο δεν απήντησαν στην έκκληση του, ε, των εμπειρογνωμόνων να αναθεωρήσουν τις οδηγίες για τις εκφράσεις μίσους ε, στο περιεχόμενο του. Το Συμβούλιο δεν δεσμεύτηκε να απεμπλέξει τις συζητήσεις για την οριζόντια οδηγία περί διακριτικής μεταχείρισης και ρατσιστικής συμπεριφοράς. Εκεί θα έπρεπε να παρέχεται σε όλου του τομεί τη ζωή, όχι μόνο στην απασχόληση, απελευθέρωση από τη διακριτική μεταχείριση λόγω σεξουαλικού, φιλετικού προσανατολισμού κτλ. Ένα αγόρι Ρωμά ε, ξυλοκοπήθηκε και προσβλήθηκε α, από άντρε που του χαρακτήρισε Ρωμά. Του είπαν. ε, ότι τι τόλμησες να πεις ότι είμαι και εγώ τσιγκάνος και τον πλάκωσαν στο ξύλο. Όλοι έμειναν άφωνοι στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Καταδίκασαν τις επιθέσεις κατά τον Ρωμά που είναι πολύ συχνά θύματα βίας και πολύ σπανιότερα δράστες. Το είπαν. Ε, ναι, α, είμαστε μαζί με τους Ρωμά στην υπεράσπιση των ανθρωπινών δικαιωμάτων τους. Πρέπει λοιπόν να είναι πιο σαφείς οι θεσμικές πολιτικές κατά του ρατσισμού και να υπάρχει συστηματικότερη χάραξή τους. Ακόμη οι πολιτικοί καιροσκόποι τις εκμεταλλεύονται. Ακούσαμε ότι είπατε αρμοστία του ΟΗΕ για τη στρεβλωμένη συζήτηση που γίνεται στην κοινή γνώμη για τους πρόσφυγες. Το πώς παρουσιάζονται πληροφορίες στον κόσμο. Και όμως μόνο ένα κράτος, ο Έλληνας εκπρόσωπος, το συνδύασε με τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το άσυλο και τη μετανάστευση που εντείνουν την τάση αυτή. Εν τέλει, ακούσαμε και έντονε μαρτυρίε για τι διακριτικέ μεταχειρήσει κατά των μουσουλμάνων, των Ισλαμιστών, λόγω τη κατάσταση έκτακτη ανάγκη στη Γαλλία. Κι όμω η νέα οδηγία για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία, που αυτή τη στιγμή είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση, δεν εγγυάται την ε, εφαρμογή και με μη διακριτικό τρόπο για τα νέα δικήματα ή που να είναι αντισυνταγματικοί ή να μην πλήττουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πράγματι και σίγουρα δεν μπορούν όλα να επιληθούν ταυτόχρονα και όλα μαζί. Στατηγική δράση πρέπει να, υπάρξει και να επικεντρωθεί στις πρώτες προτεραιότητες. Είναι σαφές. Όμως αυτή τη στιγμή, χωρίς καμία πηξίδα, με τέτοιες έκτατες ανάγκες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάπου πρέπει να βρεθεί μέση λύση μεταξύ ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών που έχουν την ετικέτα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτή η ομάδα υψηλού επίπεδου από τη μια, και από την άλλη με τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ πολιτικέ, ιδίω στον τομέα τη δικαιοσύνη και των ε, εσωτερικών υποθέσεων. Τα άρθρα 1 και 6 των συνθηκών ευαγγελίζονται τι θεμελιώδει αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω θεμέλια τη οικοδόμηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα πρόγραμμα στρατηγικό για συνοχή στι δράσει τη με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλε τι πολιτικέ τη, από το πρώτο στάδιο μέχρι την υλοποίηση και την επιβολή. Όπω πλησιάζουμε στην ενδιάμεση αναθεώρηση τη νέα Επιτροπή, και ο κύριος Τίμερμανς ε, μπορεί να, ε, θα πρέπει να δικαιολογήσει τη θέση του, νομίζω ότι καλό θα ήταν να έρθει στο κοινοβούλιο σας και να προτείνει ένα τέτοιο πλαίσιο. <clears throat> Ε, Ευχαριστώ πολύ την κυρία Καζίνσκι για την επικοδομητική παρουσίαση. Τώρα έχουμε χρόνο για κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις. Μια συζήτηση Ένας είναι ο Ευρωβουλευτής που θέλει να πάρει το λόγο, ο κύριος Σόγκο. Ευχαριστώ. Είναι περισσότερο ένα σχόλιο από αυτό που θέλω να κάνω για την πρώτη παρουσίαση της κυρίας Μαλαφ. Ένα μόνιμο πρόβλημα που έχουμε είναι πώς να πείσουμε τα θεσμικά όργανα για μια στρατηγική που ήδη υπάρχει. Υπάρχει μία έκθεση για τις εθνικές, ε, εθνοτικές ε, ε, μειονότητες και δεν θέλω να τη συγκρίνω με τους Ρωμά και να πω ότι είναι σε καλύτερη μοίρα ή χειρότερη. Έχω μόνο μία πρόταση εδώ από το αντίστοιχο έγγραφο του Κοινοβουλίου που έχει να κάνει με το σχόλιο σας που λέει ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση ε, για τον ε, χάρτη, για τις περιφερειακές ε, γλώσσες κτλ. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί το δυναμικό της νέας νομοθεσίας συστηματικά ως τώρα και δεν έχουν εφαρμοστεί οι αξίες του, της σύμβασης του Συμβουλίου για τις εθνικές μειονότητες, κυρίως λόγω της λανθασμένης αντίληψης ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες για να νομοθετήσει για τις ε, εθνικές μειονότητες. Δεν χρειάζεται αν ζητήσουμε από την Κομισιόν να φτιάξει μια λίστα με τη νομική βάση, βάση της οποίας θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, θα ήταν ένα πρώτο βήμα για την εφαρμογή του ψηφίσματος που ενέκρινε το Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2015. Ίσως γι' αυτό το λόγο δεν ήρθε ο κύριος Τίμερμανς εδώ, γιατί από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα δεν ήταν μεγάλο το διάστημα για να μπορεί να μας παρουσιάσει αυτό το έγγραφο. Ίσως ε, το καλοκαίρι ή και του χρόνου να έχουμε το έγγραφο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνταχθώ με τον ε, προλαλήσαντα σχετικά με τις εθνικές μειονότητες σε πολλά μέρη αυτής της Υπήρου υπάρχει αυτό το ζήτημα εδώ και 100 χρόνια και παραπάνω. Έχει ήδη αναγνωριστεί στο δίκαιο. Κάποιες φορές όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα δεν μπορούν να αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν το θέμα. Η κατάσταση είναι παράλογη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνήθως αναφέρεται σε αυτά τα θέματα ως εσωτερικά ε, χώρια θέματα. Όμως μιλάμε για παραδοσιακές μειονότητες. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να αποφασίζονται βάσει ε, της ε, ε, εγγενούς ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας κτλ. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε ασαφείς όρους για τις μειονότητες. Ακόμα και αν είχαμε, έχουμε μια μειονοτική γνώμη, δεν σημαίνει ότι η γνώμη αυτή είναι σωστή. Ο καθένας έχει την άποψή του. Όμως το να λέμε ότι η πολύγαμη είναι μειονότητα είναι σαν να έχουμε μία περίεργη άποψη για την ίση μεταχείριση ε, μιας οικογένειας. Ε, η μονογαμική οικογένεια είναι η βάση για το σεβασμό των γυναικών στην Ευρώπη. Είναι ένας θεσμός κλειδί που δείχνει την ισότητα ε, στην κοινωνία μας. Και γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίζουμε έτσι την πολυγαμία. Παρόλο που υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που έρχονται στην Ευρώπη και έχουν επιστοποιητικό γάμο που λέει ότι είναι παντρεμένοι με πολλά άτομα. Εμείς δεν χρειάζεται αυτό να το εφαρμόσουμε στη δική μας ένομη τάξη. Έχουμε το δικαίωμα να περασπιστούμε τα στοιχεία της κουλτούρας μας που θεωρούνται οικονομικά. Δεν οικουμενικά, δεν είναι απαραίτητα μειονοτικά. Άρα Ας μην θεωρούμε ότι κάθε μειονότητα είναι ε, ειδική και προνομιούχος. Ας μην δώσουμε συγκεκριμένα προνομιακά δικαιώματα. Να ευχαριστήσω τον κύριο ε, Μπλεκ για αυτά που είπε για τα παιδιά με σύνδρομο Down. Η κατάσταση είναι δραματική. Σε πολλά από τα κράτη-μέλη και δυστυχώς και στην Πολωνία, το δικαίωμα αυτών των παιδιών να γεννηθούν αμφισβητείται. Γιατί είναι θύματα του εγκλήματος της άμβλωσης λόγω της αναπηρία τους. Και όταν επιβιώνουν αντιμετωπίζονται ας, ως αναξιοπρεπή και κρίνονται συνεχώς από τους γονείς τους για παράδειγμα που αποφασίζουν αν τα παιδιά αυτά ε, πληρούν τις προσδοκίες τους ή όχι. Αυτό είναι απάνθρωπο κατά τη γνώμη μου. Ξέρω ότι αυτή η δήλωση βέβαια δεν θα αλλάξει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως δεν πρέπει να είμαστε ήσυχοι και όταν κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί πολλά κράτη-μέλη έχουν αποφασίσει ότι υπάρχει το δικαίωμα της απόφασης ε, όσον αφορά το δικαίωμα ενός παιδιού να γεννηθεί. Ε, δεν πρέπει να είναι μια αυθαίρετη απόφαση. Νομίζω ότι και σε αυτό το τομέα πρέπει να δούμε τα στάνταρντ, τα πρότυπα που εμείς υπερασπιζόμαστε και το πώς τα ορίζουμε. Πώς ορίζουμε επίσης την κατάσταση αυτή. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε καλύτερα το γεγονός ότι η μειονοτική άποψη δεν είναι πάντοτε η σωστή ή δεν έχει πάντοτε ισχύ, γιατί πολύ συχνά μιλάμε για μειονότητες ε, οι οποίες έχουν την ισχυρή ε, προστασία από την πλειονότητα, αλλά οι πραγματικές μειονότητες μένουν μόνες τους και σιωπούν. Ευχαριστώ. Τέλος, να πω κι εγώ κάτι ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οπότε θα ε, μιλήσω πολωνικά. Ε, ε, Ευχαριστώ. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα θέμα. Μειονότητα, η οποία παραμένει μειονότητα, βρίσκεται πάντα σε πιο δύσκολη κατάσταση από ότι μια πλειοψηφία. Ας σκεφτούμε τη, μια οικογένεια, δύο κόρες, μία μεγαλύτερη, μία πολύ μικρότερη. Πάντα η μικρότερη χρειάζεται περισσότερη προσοχή, περισσότερη φροντίδα μέχρι να έχει μεγαλώσει μέχρι να έχει φτάσει σε οριμότητα και να είναι ανεξάρτητη. Το ίδιο ισχύει και με τις μειονότητες. μπορούμε να έχουμε άπειρες συζητήσει εδώ, αλλά μην ξεχνάμε ότι οποιαδήποτε μειονότητα, είτε πρόκειται για τα άτομα με αναπηρίες, είτε μια άλλη μειονότητα, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερη φροντίδα. Και γι' αυτό και μιλήσαμε για τις μειονότητες σε αυτή τη συζήτηση και δεν είναι και η τελευταία φορά που το κάνουμε. Αυτά. Καλώς. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παρέμβει στην ε, συζήτησή μας από ό,τι έχω καταλάβει. Σύναβα Μπούκαρτ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Προς ενημέρωσή σας για τον κύριο Πατ Κλάρκ. Φυσικά και συμμερίζεται τις ανησυχίες σας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα διευθυντικά ταμεία, τα οποία πρέπει να δαπανώνται βάσει των ρυθμίσεων για τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι κι αλλιώς η ευθύνη είναι επιμερισμένη. Είναι επιμερισμένη δηλαδή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Ελέγχει τους ελέγχους που κάνουν οι χώρε μέλη η Κομισιόν. Αυτό είναι αλήθεια. Και Προς πληροφορία σας θέλω να πω ότι τον Ιούλιο ένα ερμηνευτικό κείμενο θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την διαχείριση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων σε σχέση με την Σύμβαση μελιωδών Δικαιωμάτων. Θα εγκριθεί αυτό το ερμηνευτικό κείμενο λοιπόν και από εκεί και πέρα περιμένουμε και από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις στις χώρες μέλη να μας ενημερώνουν και να μας βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση για αυτά τα θέματα. Δεύτερον, για την κυρία Κωνσασκίνα. Πολύ καλά τονίσατε ότι στην ετήσια έκθεση όταν αναφερόμαστε στις διαδικασίες προσφυγής μερικές φορές κατανομάζουμε τις χώρες μέλη που κάνουν παραβιάσεις, άλλες φορές όχι. Παρ' αυτά, παρόλο που μπορεί να μην φαίνεται εκ πρώτης άψεως, υπάρχει κάποια συνοχή κάθε φορά που υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαδικασίες επί παραβάση και όπου κατανομάζεται τότε κάποια χώρα, τότε και στην ετήσια έκθεση αναφέρεται αυτό. Για τις διαδικασίες επί παραβάση όμως, όπου δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση ή ε, δηλώση στον τύπο, τότε δεν αναφέρεται η ε στον τυπο τοτε ούτε στην ετήσια έκθεση. Ελπίζω να διευκρίνησα έτσι κάπως τα πράγματα σε ευχαριστούμε. Τώρα, φαντάζομαι ότι θέλετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις, έτσι. Παρακαλώ, εσείς πρώτα. Προς τον κύριο Σόγκαρ, λέει η κυρία Μαλόη, θέλω να πω ότι αναφέρατε την ετήσια έκθεση για τις μειονότητες. Εμείς βασιζόμαστε στην Γερμανία, σε μια περιοχή της Γερμανίας και η τοπική εκεί η αρχή κάθε χρόνο έχει αιτήσει έκθεση για τις μειονότητες που αναγνωρίζει η Γερμανία. Τρεις από αυτές βρίσκονται και στην περιοχή σε μεγάλο αριθμό. Και είναι μια κοινή προσπάθεια, έτσι δεν είναι κάτι που γράφουν από μόνοι τους οι και οι οργανώσει, οργανώσεις, κοινωνία των πολιτών συμμετέχει. Όσον αφορά τι αρμοδιότητες, αναφερθήκατε σε μια έκθεση που βεβαίω. Κυρίως όταν πρόκειται για ουσιαστικά δικαιώματα σχετικά με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό και ο κύριος Τη είπε. Στον κύριο Γκρέκ θέλω να πω ότι ένα από τα πολιτιστικά αυτά δικαιώματα θα μπορούσε να το ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να το υποστηρίξει ως ένα οικουμενικό δικαίωμα. Γιατί όλα τα μέλη της κοινωνίας λένε ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν είχα καιρό να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πολλές χώρες που παρακολουθούμε, υπάρχει και στην έκθεση που σας έδωσα, στη γραμματεία, είναι θέμα ανησυχίας πώς μεταγράφεται το όνομα και πρέπει την ταυτότητά τους όντως οι μειονότητες να μπορούν να τη διατηρήσουν όπως και τη γλώσσα τους και τον πολιτισμό τους. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να κάνει κάτι και να το συμπεριλάβει για να εφαρμόσει περισσότερο ουσιαστικά δικαιώματα των μειονοτήτων. Θέλω επίσης να πω ότι το κατά πόσο μια άποψη μειονότητας είναι σωστή ή λάθος, αυτό φυσικά είναι υποκειμενικό σας υπενθυμίζω όμως ότι είναι σημαντικό να ακούγεται κάθε φωνή στη δημοκρατία. Είτε είναι σωστή είτε είναι λάθος. Από εκεί και πέρα, αν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, αυτό είναι άλλο. Αλλά όλοι οι δύο δι πρέπει να είναι ανοιχτοί, ώστε να ακούγονται όλες οι φωνές. Δεν σημαίνει ότι κερδίζει ο ένας ή ο άλλος, αλλά όλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν σε ευχαριστούμε. Πολύ καλό συμπέρασμα τη συζήτηση αυτό. Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ όλους τους ομιλητές για τις τόσο ενδιαφέρουσες εισηγήσεις σας και τα σχόλιά σας. Όντως, αυτά που ακούσαμε μας εμπνέουν στο έργο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους.